and gentlemen. Καλή σας ημέρα. Παρακαλώ καθίστε. Thank you Ευχαριστώ τους παρόντες. Ευχαριστώ τα μέλη της Επιτροπής μας ε, που έφτασαν εγκαίρως για τη συνεδρίαση της Επιτροπής. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας με την έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Έχω κάποια σχόλια επ' αυτής. Έχω λάβει το αίτημα από τον κύριο στην Ρόι για προσθήκη στην ημερήσια διάταξη. Αυτή η προσθήκη αφορά το σχέδιο ψηφίσματος που ακολουθεί μια προφορική ερώτηση σύμφωνα με τον κανονισμό 128 για το ζήτημα της εφαρμογής της πολιτικής συνοχής. Το κείμενο αυτού του σχεδίου ψηφίσματος σας έχει σταλεί από χθε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και προτείνω να το εξετάσουμε στο τέλος της απογευματινής μας συνεδρίασης. μια που ως τελευταίο ουσιαστικό θέμα για την Μισή Διάταξη πριν από τις ενέργειες των συντονιστών. Έτσι θα έχουμε την ευκαιρία να λάβουμε υπόψη μας τις προφορίες που πρόκειται να λάβουμε από την Επίτροπο συμπεριλαμβανομένης και αυτής της ε, ενημέρωσης περί του σχεδίου ψηφίσματος. Ε, γίνεται αποδεκτή η πρόταση αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Οπότε με αυτό το επιπρόσθετο σημείο στην ημερήσια διάταξη υποθέτω ότι μπορούμε να την εγκρίνουμε. Να συνεχίσουμε τώρα με τις ανακοινώσεις της Προέδρου. Δεν έχω καμία ανακοίνωση για σήμερα. Ίσως στο τέλος της συνεδρίασης να έχουμε κάτι να μοιραστούμε μαζί σας. Να συνεχίσουμε λοιπόν με το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, ε, εργαστήριο για τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες. Ε, ζητήθηκε από το ερευνητικό τμήμα που υποστηρίζει το, τη δουλειά της Επιτροπής μας, ε, το τμήμα πολιτικής ε, Β, το θεματικό τμήμα Β, να ασχοληθούμε με το θέμα αυτό και όπως είδατε και από το πρόγραμμα θα ε, συζητήσουμε με εμπειρογνώμονες διάφορα σχετικά θέματα θα ξεκινήσουμε με τις παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών μας και μετά θα συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψεων και τις ε, ερωταποκρίσεις με τα μέλη της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Έχουμε χρόνο για το σημείο αυτό της ημερήσιας διάταξης ως τις 11 η ώρα το πρωί ε, τότε περιμένουμε την Επίτροπο, ε, την κυρία ε, Κρέντου, να έρθει να ανταλλάξει απόψεις μαζί μας. Χωρίς να χρονοτριβώ άλλο, να δώσω το λόγο στην Ντοροτέα Λέν και στον καθηγητή Σπαν, τον Ντέιβι Σκόρνα που είναι ο γενικός ο διευθυντής που είναι υπεύθυνος για ε, τα θέματα αυτά και ε, τον ε, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Τσεχικής Δημοκρατίας. Κυρία Ντυπρέ, μήπως θέλετε να αρχίσετε εσείς. Ευχαριστώ. Εγώ είμαι η Ντοροτέα Λέντιπρέ από τον Σα ε, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να συμμετάσχω στο σημερινό εργαστήριο. Θα σας πω ορισμένα πράγματα για την αποτελεσματική δημόσια επένδυση σε υποεθνικό επίπεδο σε ε, περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών. Δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, η σημασία της διάστασης της διακυβέρνησης ε, για την αποτελεσματική δημόσια επένδυση και ε, η χρήση των ερεσιμοτήτων ως ένα παράδειγμα ε, εργαλείου διακυβέρνησης, ενίσχυσης ε, μιας μεγάλης επένδυσης. Θα ήθελα καταρχάς να σας πω μερικά γενικότερα πράγματα για το τι σημαίνει ακριβώς για τον ε, ΟΣΑ το θέμα αυτό ε, της, δημόσιας, ε, της αποτελεσματικής δημόσιας επένδυσης είναι κάτι το οποίο μπορεί να προσμετρηθεί, είναι κάτι το οποίο μπορεί να υπολογιστεί όμως εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το, τη διαχείριση της επένδυσης αυτής και τη διακυβέρνηση. Η καλή διακυβέρνηση λοιπόν της δημόσιας επένδυσης έχει άμεση σχέση με τον αντικτυπό τη και μιλούμε για τη διακυβέρνηση σε εθνικό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο υποεθνικό κυρίως. Έχουμε κάποιες εμπειρικές μελέτες που δείχνουν ότι η ποιότητα της ε, περιφερειακής διακυβέρνησης έχει άμεσο αντίκτυπο στην αποτελεσματικότητα της χρηματοδότησης και αυτό ισχύει όλος ιδιαίτερο στην περίπτωση των ταμείων συνοχής για παράδειγμα. Για ποιο λόγο λοιπόν οι υποεθνικές ε, κυβερνήσεις είναι τόσο σημαντικές για τη δημόσια επένδυση, για τι δημόσιες επενδύσεις. Γιατί ακριβώς αυτές ε, οι αυτοδιοικήσει είναι πάρα πολύ σημαντικές ε, στο μέσο όρο στι χώρε του ΩΣΑ. Είναι το 16% το, το 60% συγγνώμη, των επενδύσεων, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι το 55%. <clears throat> αν δούμε λίγο το, τη συγκυρία αυτή τη στιγμή, υπάρχει μία μείωση στη δημόσια και ιδιωτική επένδυση από τότε που ξεκίνησε η κρίση και αυτό ισχύει σε όλες τις χώρες του ΩΣΑ και πολύ περισσότερο στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης και βλέπετε εδώ στην γραφική παράσταση με το κόκκινο είναι η μείωση σε ε, δημόσιες επενδύσεις σε υποεθνικό επίπεδο στην Ευρωπαϊκή Ένωση από το 2009 και εξής. Βλέπετε ότι οι δημόσιες επενδύσεις έχουν χρησιμοποιηθεί σαν ε, ε, μεταβλητή ε, προσαρμογής μέσω, για παράδειγμα, φορολογικών δαπανών, οι οποίες έχουν αυξηθεί όμως κάναμε και μία πρόσφατη μελέτη όσον αφορά τα βασικά εμπόδια για την, ε, τις υποεθνικές δημόσιες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό που μπορούσαμε να δούμε είναι ότι τα βασικά εμπόδια στη διακυβέρνηση ε, θεωρήθηκαν τόσο σημαντικά όσο και οι ε, χρηματοοικονομικές προκλήσεις. 90% ε, των ε, ερωτηθέντων είπαν ότι οι διοικητικές διαδικασίες είναι πάρα πολύ μακροχρόνιες, ότι υπάρχει γραφειοκρατία και ότι αυτές είναι μεταξύ των βασικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η δημόσια επένδυση. Επίσης αναφέρθηκε η έλλειψη ικανότητας ε, προγραμματισμένη στρατηγικής δημόσιας επένδυσης ε, μακροχρόνια, όπως επίσης το γεγονός ότι ο συντονισμός ε, μεταξύ των τομέων και μεταξύ των διαφόρων επιπέδων της κυβέρνησης δεν ήταν ο σωστός. Υπάρχουν επίσης ε, και ε, και καλές πρακτικές οι οποίες ε, έχουν αρχίσει να ισχύουν σε υποεθνικό επίπεδο και μπορούμε να δούμε από την έρευνά μας την περσινή ότι είναι αρκετές αυτές οι προσπάθειες. Όσον αφορά τη γενική σύσταση που θα μπορούσαμε να κάνουμε για εθνικό και υποεθνικό επίπεδο ως προς τις κυβερνήσεις δηλαδή για την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων μπορούμε να δώσουμε ορισμένα ορισμένες, ε, να κάνουμε τις εξής συστάσεις. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα, ένας μεσοπρόθεσμος προγραμματισμός, ε, να υπάρχει ανάπτυξη πολιετούς ε, προϋπολογισμού, και για την εθνική, και τις εθνικές κυβερνήσεις είναι ουσιώδες να υπάρξουν κίνητρα προκειμένου να συμμετέχει και να συνεργάζεται σε, κοινές, σε κοινά επενδυτικά, δημόσια επενδυτικά προγράμματα και η κυβέρνηση σε υποεθνικό επίπεδο. Έχουμε ένα νομικό ε, μέσο ε, το οποίο εγκρίθηκε από 35 χώρες του ΩΣΑ ε, υπάρχουν εκεί κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, κάποιες αρχές για το πώς τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης πρέπει να διαχειριστούν τις δημόσιες επενδύσεις με συντονισμένο τρόπο και επίσης ε, παρακολουθούμε το βαθμό στον οποίο τα κράτη-μέλη και οι υποεθνικές κυβερνήσεις ε, εφαρμόζουν το συγκεκριμένο νομοθετικό μέσο. Έχουμε λοιπόν στον ιστότοπό μας ένα kit ένα πακέτο εργαλείων εφαρμογής με καλούς δείκτες για το πώς τα διάφορα επίπεδα της κυβέρνησης μπορούν ε, ή θα έπρεπε να ε, διαχειρίζονται τις δημόσιες επενδύσεις. Αν επικεντρωθούμε τώρα στα συγκεκριμένα από παραδείγματα της χρήσης των ερεσιμοτήτων, ε, ένα παράδειγμα ε, ενό μέσου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της χρηματοδότησης. Είναι ε, ένα πολύ, μια πολύ ευρία έννοια η έννοια της αιρεσιμότητας γιατί Πρόκειται για ένα στοιχείο οποιασδήποτε χρηματοοικονομικής ε, μεταφοράς που δεν είναι ένα καθαρό δώρο. Υπάρχουν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες οι οποίες πρέπει να πληρούνται εκ των προτέρων ε, πριν από κάθε συμβατική ε, υποχρέωση, πριν από κάθε, την υπογραφή κάθε σύμβασης. Αν επικεντρωθούμε περισσότερο στην εμπειρία από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Παγκόσμια Τράπεζα, που ε, βεβαίως είναι πολύ γνωστά για τη χρήση των αιρεσιμοτήτων ε, εδώ και δεκαετίες, υπάρχουν κάποια διδάγματα τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε. Υπάρχει σημαντική αύξηση της χρήσης των αιρεσιμοτήτων ε, στη δεκαετία του 80 και του 90 αλλά έχει έχουν υπάρξει και επικρίσεις ε, εναντίον τους ότι δεν ήταν αποτελεσματικές όσον αφορά την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της κοινωνικής ευημερίας. Ε, κάποια από τις επικρίσεις αφορούσε το ότι όταν υπάρχουν πάρα πολλοί λεπτομερείς ε, όροι που ισχύουν, τότε είναι πάρα πολύ χρονοβόρο να γίνουν οι διαπραγματεύσεις, υπάρχουν και αντιφάσεις. Έχουν γίνει λοιπόν κάποιες αλλαγές κατά τη δεκαετία του 2000. Ο στόχος ήταν η μείωση του αριθμού των ερεσιμοτήτων που ισχύουν ε, για να υπάρξει περισσότερη ευελιξία στον τρόπο με τον οποίο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έρχεται σε επαφή με τις χώρες και εμπλέκεται στις χώρες αυτές ε, ως προς τις μεταρρυθμίσεις ε, υποτίθεται ότι τώρα οι αιρεσιμότητες είναι καλύτερα προσαρμοσμένες ε, στις ανάγκες των χωρών, λιγότερο αυστηρές και υπάρχει μεγαλύτερη εστίαση στις ε, κυβερνήσεις και στα θεσμικά κριτήρια όπως επίσης και σε περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα. Και η Παγκόσμια Τράπεζα εστιάζει λίγο περισσότερο στις ε, εκ των υστέρων Όλες οι χώρες του ΩΣΑ βεβαίως ε, χρησιμοποιούν κάποιου είδους αιρεσιμότητες όταν χρησιμοποιούν ε, επιδοτήσεις για ε, σε επίπεδο υποεθνικής αυτοδιοίκησης, τουλάχιστον για την περιφερειακή ανάπτυξη, σε 20 χώρες αφορά ε, τους ε, τομείς, τα ταμεία δημοσίων ε, επενδύσεων, επενδύσεων που χορηγούνται από τις εθνικές κυβερνήσεις. Βλέπετε λοιπόν κάποιες κάποιοι όροι που πρέπει να ισχύουν όσον αφορά στο χρονοδιάγραμμα, για παράδειγμα, όσον αφορά την ε, πρικοδότηση συγκεκριμένων στόχων για την εφαρμογή των αιρεσιμοτήτων αυτών. Κάποια ε, διδάγματα τώρα από την διεθνή εμπειρία ως προς τις αιρεσιμότητες ε, από μόνες τους πολύ σπάνια ε, αρκούν για να υπάρξει πραγματική αλλαγή που θα διαρκέσει στο χρόνο. Δεν πρέπει να είναι πολύ περιοριστικές, πρέπει να συνοδεύονται από σημαντική τοπική ηγεσία και πολιτική υποστήριξη ε, πρέπει να, μπορούν, να, να μπορούμε να τις παρακολουθήσουμε η αξιοπιστία του συστήματος είναι πάρα πολύ σημαντική. Χρειάζονται μηχανισμοί επιβολής βεβαίως ε, και μία αξιόπιστη ικανότητα από το υψηλότερο επίπεδο το, της κυβέρνησης να παρακολουθούν την αποτελεσματική εφαρμογή. Και κάτι ακόμη ε, το να εστιάζουμε ε, στα, ε, ε, στο αποτέλεσμα και στην ανταμοιβή πιο εύκολα θα λειτουργήσει από ότι η σκέτη όρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες στον ιστότοπό μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σπάν, θα θέλατε να συνεχίσετε. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Μιχαήλωβα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Με χαρά μου θα σας παρουσιάσω την έρευνα για την αρεσιμότητα στα διακυβερνητικά δάνεια, εξετάζοντας την περίπτωση των Ηνωμένων Πολιτειών και συγκρίνοντάς την με την κατάσταση εδώ στην Ευρώπη. This the right button to press. The right button, okay. Uh, my presentation... Η παρουσίασή μου θα χωρίσει σε τέσσερα τμήματα. Ε, καταρχάς, τι είναι μια επιχορήγηση υπό προϋποθέσεις. Η αιρεσιμότητα έχει διάφορες πτυχές. Έπειτα θα κοιτάξουμε τα ομοσπονδιακά ε, τις ομοσπονδιακές επιχορηγήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών και τα προγράμματα σχετικά, μετά τις ε, συγκρίσεις με την ευρωπαϊκή φιλοσοφία και τις, θα εξετάσουμε την ε, αιρεσιμότητα στην περιφερειακή πολιτική. Καταρχάς πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός ανάμεσα στις γενικέ αρχές οι οποίες χρειάζονται για να ε, εξασφαλίσουμε χρηστή διακυβέρνηση και ισότητα και ε, να δούμε την αισθήση σε στρατηγικούς στόχους. Όταν ε, προετοιμάζεσαι για ένα έργο πρέπει να έχεις ένα συγκεκριμένο πλάνο, ένα στόχο. Διαφορετικά δεν μπορείς να λάβεις επιχορήγηση. Μετά υπάρχουν διάφορες προποθέσει θεματικού τύπου. Καταρχάς, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα πολιτικών και οι προτεραιότητες πολιτικής να μπορούν να υιοθετηθούν από τις κυβερνήσεις που λαμβάνουν τις ε, επιχορηγήσεις. Είναι ένα αρκετά αμφιλεγόμενο θέμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι αυτό σημαίνει ότι οι Βρυξέλλες ε, ορίζουν τις δικές τους ε, προτεραιότητες στις κυβερνήσεις των κρατών μελών. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα αρκετά λεπτό ζήτημα. Εάν δούμε το πλαίσιο του κανονισμού 1303, Έχουμε τις γενικές προϋποθέσεις ε, για την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα. Υπάρχουν 29 ε, θεματικές προϋποθέσεις και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δεν εμφανίζονται καν στο πρώτο κομμάτι του κανονισμού. Εμφανίζονται στη συνέχεια, όταν δηλαδή δεν διαβάζουν πλέον οι πολιτικοί, έχουν σταματήσει να διαβάζουν τον, να τον κανονισμό. Αναφέρονται σε συγκεκριμένους στόχους και την επίτευξη τους, ε, στόχοι που μπορεί να είναι είτε εθνικοί είτε ευρωπαϊκοί. Και αυτό είναι σημαντικό. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες οι επιχορηγήσεις δίδονται από ομοσπονδιακέ υπηρεσίες και δεν υπάρχει κάποια κεντρική αρχή. Όμως, Αυτές ε, οι επιχορηγήσεις, όπως είπα, δεν είναι συντονισμένες από κάποια κεντρική αρχή, μπορούν όμως να ταξινομηθούν με βάση κάποια γενικά επίσημα χαρακτηριστικά. Αυτό λοιπόν ονομάζεται Federal Domestic Assistance, Ομοσπονδιακή Εγχώρια Βοήθεια. αλλά δεν είναι όλα επιχορηγήσεις. Υπάρχουν διάφορες μορφές, δάνεια τύπου, άμεσα δάνεια, ασφαλίσεις και ε, υπάρχουν διάφορες ε, επιχορηγήσεις ή ενισχύσεις υποεθνικών υπηρεσιών, οι οποίες ε, δεν διέπονται από συγκεκριμένους κανόνες. Υπάρχουν περίπου 1.850 ε, προγράμματα, ονομάζονται επιχορηγήσεις κατηγορίας, χορηγούνται για συγκεκριμένο σκοπό και περίπου 1.600 για συγκεκριμένα προγράμματα. Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι αυξάνεται ο αριθμός αυτών των ε, επιχορηγήσεων οι οποίες έχουν τη μορφή συνεργατικών προγραμμάτων, συνεργατικών συμφωνιών. Αυτά τα προγράμματα είναι πολύ συγκεκριμένα, ε, είναι ε, προσαρμοσμένα στις ε, συγκεκριμένες ανάγκες της κάθε ομοσπονδιακής υπηρεσίας. Και η χρηματοδότηση εδώ, όπως βλέπετε, για το Υπουργείο Υγείας έχει ο, ε, ως Είναι πολύ μεγαλύτερη από, τις, από τα υπόλοιπα Υπουργεία. Τώρα, τι μπορούμε να δούμε από το παράδειγμα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, καταρχάς υπάρχουν πολλές ομοιότητες με την Ευρώπη. Υπάρχει η επιλεξιμότητα του υποψήφιου προς επιχορήγηση, υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες πριν από αυτή την επιχορήγηση, ανάλυση κόστους ε, όφελους, ε, περιβαλλοντικές μελέτες κτλ. Ανάλυση των υποδομών που θα διασφαλίσουν την επιτυχία του έργου και μετά υπάρχει η τήρηση των γενικότερων οικονομικών κανόνων, τυπικές προϋποθέσεις, ε, προϋποθέσεις σχετικά με τη συγχρηματοδότηση, υποχρέωση ε, για να χρησιμοποιηθούν και οι ιδιωτικοί επενδυτές, δαπάνες. Οι δαπάνες είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πτυχή, διότι δεν υπάρχουν περιορισμοί ως προς τις δαπάνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι κάτι που χρησιμοποιούν οι Ηνωμένε Πολιτείε και σημαίνει δηλαδή ότι εάν ε, δώσει χρήματα σε μια κυβέρνηση, η κυβέρνηση αυτή θα μπει στον πειρασμό να μειώσει τι δικέ τη δαπάνε για το συγκεκριμένο σκοπό, έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα συνεχίσει παρά την επιχορήγηση της προσπάθειες για ε, χρηστή διαχείριση κονδυλίων. Με τη μέθοδο αυτή η κυβέρνηση υποχρεώνει την, ε, τον δικαιούχο να ασκήσει αυτή την ε, χρηστή διακυβέρνηση. Τώρα υπάρχουν κάποιες ε, εκ των υστέρων προϋποθέσεις και υποχρέωση υποβολής εκθέσεων. Τώρα έχει ασκηθεί κριτική σε κάποια από αυτά τα προγράμματα γιατί συνοδεύονται από διοικητικό άχθος, υπάρχει επικάλυψη και υπάρχουν επίσης πολλοί περιορισμοί οι οποίοι εμποδίζουν τις επιχορηγήσεις αυτές να προσαρμοστούν στις ανάγκες της ε, συγκεκριμένης ε, περιφέρειας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την περιφερειακή πολιτική. Στην περιφερειακή πολιτική ακολουθείται μια περισσότερο γραμμική προσέγγιση. Όταν όμως δούμε την οριζόντια διάσταση της περιφερειακή πολιτική συνειδητοποιούμε τα προβλήματα που υπάρχουν. Τώρα, ε, γίνεται, γίνεται διαγωνισμός για την ε, χορήγηση μιας τέτοιας ε, ενίσχυσης. Εδώ υπάρχει διαφορά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου υπάρχει υποχρέωση δίκαιης μεταχείρισης ε, όλων, δεν αποκλείονται κάποιες ε, χώρες μόνο και μόνο επειδή δεν είναι σε θέση να διαχειριστούν σωστά την επιχορήγηση. Και, όπως σας είπα, πρέπει να επιτρέψουμε πετύχουν οι τοπικές κυβερνήσεις με τις επιχορηγήσεις αυτές συγκεκριμένους στόχους, αυτό που δεν βλέπουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για παράδειγμα, η νόμιμη ηλικία που μπορεί να πιει κάποιο αλκοόλ στις ΗΠΑ είναι τα 21 έτη, η ανώτατη ταχύτητα στις ε, εθνικές οδούς είναι 55 μίλια την ώρα. Αυτά είναι ε, αυτοί είναι στόχοι οι οποίοι έχουν τεθεί σε ομοσπονδιακό επίπεδο. Όμως οι πολιτείες, οι ομοσπονδιακές κυβερνήσεις έχουν την υποχρέωση τήρησης αυτών των στόχων, διαφορετικά δεν λαμβάνουν επιχορηγήσεις. Φανταστείτε τι θα γίνει, τι θα γινόταν μάλλον στην Ευρώπη, εάν οι Βρυξέλλες επέβαλαν στη Γερμανία ανώτατο όριο ταχύτητας. Χαμός. Εδώ λοιπόν υπάρχει αυτή η διαφορά ε, και αυτό εξηγείται με το ότι είναι, είναι προαιρετική η ε, αίτηση λήψης αυτής της επιχορήγησης. Ε, οπότε ακολουθούν το σκεπτικό ότι αν το θέλεις πρέπει να τηρείς ορισμένους κανόνες. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα πράγματα είναι διαφορετικά. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε έναν κανόνα για όλα, να ε, υπάρχει χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Αυτό σίγουρα είναι μια έννοια που για πολλούς είναι κάπως φιλοσοφική, όμως ε, στις Ηνωμένες Πολιτείες υπάρχει διαφορά, υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, δεν υπάρχει κάποιος κεντρικός συντονισμός όπως σας είπα. Τώρα, τα μέσα που υπάρχουν στη διάθεση των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως σας είπα υπάρχουν πάρα πολλά προγράμματα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως υπάρχουν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία, τα οποία ε, είναι τρόπον την ένα συντονιστικό όργανο, με ευρία έννοια. Ακριβώς γιατί η κανόνες είναι ε, παρεμφερείς. Επίσης υπάρχουν και εξαιρέσεις όπως θα γνωρίζετε. Τώρα, αν δούμε τις κεφαλιακές επιχορηγήσεις, θα δούμε ότι ε, στις Ηνωμένε Πολιτείε είναι γενικότερος ε, γενικότερη η στόχη, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν λαμβάνεται μια επιχορήγηση έτσι γενικά. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένος σκοπός η επιχορήγηση να διατεθεί για συγκεκριμένο σκοπό. Επίσης, οι Ηνωμένε Πολιτείες ε, καταβάλουν πληρωμές σε ε, άτομα. Για παράδειγμα, με τα προγράμματα Medicaid, Medicare. Αυτό είναι ένας στόχος πολιτικής της Ομοσπονδιακής κυβέρνηση. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση όμως δεν υπάρχει κάποια ε, πολιτική κοινωνική πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο για όλους. Οι πολιτικές αυτές είναι έμεσες μέσω των ε, εθνικών κυβερνήσεων. Τώρα υπάρχουν συγκεκριμένα κεφα... συγκεκριμένες κεφαλαϊκές επιχορηγήσεις στις Ηνωμένε Πολιτείες, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση όχι παρά το γεγονός ότι στα διαρθρωτικά ταμεία δίδεται έμφαση στην ε, ανάπτυξη και στις επενδύσεις. Το σχέδιο Γιούνκερ, παράδειγμα. Τώρα υπάρχουν ορισμένες προκλήσεις. Ε, ας ε, δούμε τις Ηνωμένε Πολιτείε λίγο σύντομα. Υπάρχει βέβαια ένα πρόβλημα συνοχής της στρατηγικής το οποίο υπάρχει εν μέρει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα μέσα αυτά πρέπει να συνδέονται με, την, ε, με τις διάφορες στρατηγικές, από την Ευρώπη 2020 κτλ. Μετά προσπαθούμε να βελτιστοποιήσουμε τις ε, συνέργειες των διαρθρωτικών επενδύσεων. Και το βασικό ερώτημα είναι το εξής. Πρέπει να επιβραβεύουμε ή να τιμωρούμε τις ε, καλές ή άσχημες επιδόσεις αντίστοιχα. Μετά, απλοποίηση των κανόνων υλοποίησης ε, είναι μια πρόκληση και χρειάζεται βελτίωση στους ε, ελέγχους του αποτελέσματος. Χρειάζεται να κοιτάξουμε δηλαδή το αποτέλεσμα και όχι τα ε, κριτήρια εκ των προτέρων. Τώρα, βέλτιστες πρακτικές. είναι ενδιαφέρον αυτό που κάνουν οι Ηνωμένε Πολιτείε. Προσπαθούν να συνδέσουν διάφορα έργα ε, με, ε, με επιχορηγήσεις ε, μπλοκ, συνολικές. Προσπαθούν να συνδέσουν λοιπόν προγράμματα υπό συγκεκριμένες γενικές προϋποθέσεις και έτσι λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι επιχορηγήσεις σε μπλοκ. Για παράδειγμα, η ενίσχυση στα εξαρτώμενα μέλη μιας οικογένειας, παιδιά. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την άλλη, υπάρχει μια στρατηγική διπολιτική συνοχής, υπάρχουν ε, ρυθμιστικές και θεσμικές προϋποθέσεις, οι οποίες διέπουν αυτές τις ε, επιχορηγήσεις. Επίσης υπάρχει ενίσχυση της συγχρηματοδότησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα κράτη-μέλη συμμετέχουν ενεργά στην διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό να είναι επιτυχημένα ε, τα προγράμματα που λαμβάνουν επιχορηγήσεις. Μετά, από κοινού διαχείριση και έλεγχος ε, των διαρθρωτικών ταμείων. Εδώ να πω ότι αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα που έχουμε σε σχέση με τις Ηνωμένε Πολιτείε, οι οποίες δεν διαθέτουν ένα τέτοιο μέσο και μετά ε, μόχλευση σχετικά με τα δάνεια, υποχρέωση για ιδιωτικέ επενδύσει κτλ. Τώρα, οι συνολικές προποθέσει έχουν κάποιες λεπτομέρειες τις οποίες αξίζει να εξετάσουμε. Υπάρχουν λοιπόν μερικές γενικές προϋποθέσεις που ταξινομούνται κατά τύπο, κατά θέμα. Το πρόβλημα είναι να αποφασίσει κανείς εάν κάτι είναι επιλέξιμο ή όχι. Αυτό το ερώτημα δεν ε, υφίσταται στις Ηνωμένε Πολιτείε, ακριβώς γιατί οι επιχορηγήσεις δίδονται για συγκεκριμένο σκοπό. Ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν κάποια κριτήρια γενικότερα και αν ένα ε, έργο, μια πρόταση πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, ε, εφαρμόζονται τα κριτήρια, μπορεί να ε, χορηγηθεί επιχορήγηση. Ορισμένες ε, προϋποθέσεις όμως ε, είναι μόνο στο χαρτί. Δηλαδή, για παράδειγμα, ζητήματα που αφορούν την ισότητα των φύλων. Πολλές φορές το να πάρεις μια επιχορήγηση ή όχι εξαρτάται αν θα, ε, συμπληρώσεις το κουτάκι για ε, την ισότητα, ας πούμε. Και μπαίνει σε πειρασμό να το κάνεις παρότι δεν ε, έχεις προβλέψει κάτι τέτοιο στο, στην πρότασή σου. Εδώ αναφέραμε επίσης την ε, υλοποίηση των προϋποθέσεων και βρήκα μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση ότι, ότι τα κράτη-μέλη θεωρούν σε γενικές γραμμές την εκ των προτέρων αιρεσιμότητα ως ε, επιλέξιμη και δέχονται αυτε, ότι αυτές οι προϋποθέσεις ε, μπορούν να υλοποιηθούν. Τώρα, βλέπουμε εδώ αυτές τις περιπτώσεις ε, στον οριζόντιο άξονα έχουμε ε, τη θεματική επιλεξιμότητα και βλέπουμε αν μπορεί να εφαρμοστεί. Ναι ή όχι. Στην αρχή του γραφήματος βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές ε, που είναι σχετικές όμως και ακόμα περισσότερες οι οποίες είναι κάτω από το 8% και δεν είναι σχετικές με την ε, κάθε περίπτωση. Στις Ηνωμένες Πολιτείες αυτές οι περιπτώσεις ε, ούτε καν θα ε, εξετάζονταν ως υποψήφιες. Μετά, ας αναλύσουμε αυτή τη μία εφαρμογή, θα δούμε ότι το 10% είναι οι περιπτώσεις οι οποίες δεν είναι υλοποιήσιμες. Μετά, 22% μάλλον 68% ε, το κίτρινο κομμάτι είναι περιπτώσεις που θεωρούνται μη εφαρμοστές, όμως ε, σε γενικές γραμμές είναι εντάξει και το 22% είναι ένα γενικό και όριστο όχι. Τώρα, εάν εξετάσουμε τις προϋποθέσεις των επιχορηγήσεων για την περιφερειακή πολιτική, θα δούμε ότι στις Ηνωμένε Πολιτείε ε, είναι πολύ συγκεκριμένες και αυτό είναι κάτι στο οποίο ασκείται κριτική. Για παράδειγμα, μόνο 3% των επιχορηγήσεων κατηγορίας πηγαίνουν στην περιφερειακή ανάπτυξη. Βέβαια, η γενικότερες προϋποθέσεις πιστεύω πως δεν είναι κατάλληλες στην περίπτωση της περιφερειακής ανάπτυξης, ακριβώς γιατί χρειάζονται προσαρμοσμένες προϋποθέσεις για την κάθε περιφέρεια. Δεν, δεν είναι κάτι που πρέπει να αγνοούμε, γιατί αντιτίθεται στην ίδια τη φιλοσοφία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, χρειάζεται συνέπεια με μια περιφερειακή στρατηγική και αυτό πρέπει να είναι προϋπόθεση. Αυτό δεν μπορούμε να το βρούμε προς το παρόν στην αιρεσιμότητα. Χρειάζεται λοιπόν η κυβέρνηση να έχει συγκεκριμένο σχέδιο στρατηγικής για μια περιφέρεια. Και μετά μπορείς να προσαρμόσεις το σύστημα των επιχορηγήσεων σύμφωνα με αυτές τις ε, συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες προϋποθέσεις. Μετά χρειάζεται μια πολυδιάστατη πολυτομεακή πολιτική, διότι αυτό αποτρέπει το, την περίπτωση χρηματοδότησης έργων τα οποία δεν μπορούν να εφαρμοστούν γενικότερα. Δεν μπορούμε να αντλήσουμε όλα τα ωφέλη. Μετά, χρειάζεται φυσικά συνεργασία ανάμεσα σε, όλε, σε όλους τους ενδιαφερόμενους ε, φορείς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι σε αυτόν τον τομέα οι Ηνωμένε Πολιτείες είναι πολύ πιο ευέλικτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο τρόπο ε, με τον οποίο λειτουργούν έχει κάποια συγκριτικά πλεονεκτήματα, παρά το γεγονό ότι μόνο το 3% των επιχορηγήσεων πηγαίνει σε περιφερειακή ανάπτυξη. Τώρα, ε, διασυνοριακή συνεργασία. Α δούμε αυτήν την τυχή. Όταν ε, εξετάζουμε μια περιφέρεια, φυσικά δεν σταματάμε στα εθνικά σύνορα. Περνάμε σε διασυνοριακά ζητήματα. Και εδώ μπορεί να παρουσιαστεί ένα μικρό πρόβλημα, διότι η περιφερειακή πολιτική ιδανικά θα έπρεπε να επενδύει σε ένα περιφερειακό κέντρο ανάπτυξης ή τα χρήματα να ε, διατεθούν, να διασκορπιστούν με βάση την αρχή της δίκαιης ανταπόδοσης. Χρειάζεται λοιπόν μια ισορροπία. Ιδιαίτερα εμείς που ζούμε στις Βρυξέλλες, στο Βέλγιο, ξέρουμε πολύ καλά πόσο σημαντική είναι η ισορροπία και η διατήρησή της στην περιφερειακή πολιτική. Αυτά από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και θα χαρώ να απαντήσω σε ερωτήσεις. Ευχαριστώ κύριε καθηγητά για την ενδιαφέρουσα αυτή προσέγγιση. Ο κύριος Μπέρκοβιτς έχει το λόγο για να δούμε κατά πόσο συμφωνεί με αυτά τα ευρήματα. Ευχαριστώ. Καταρχάς να εκφράσω την ικανοποίηση που βρίσκομαι σήμερα εδώ για να παρουσιάσω την μελέτη. Φυσικά η Επιτροπή σας εμπλέκεται, μάλλον η Επιτροπή ασχολήθηκε εδώ και καιρό με το ζήτημα και νομίζω ότι είναι ένα θέμα που έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά για την ερεστιμότητα εξάνεται, ειδικά όταν συγκρίνουμε την, με τις ΗΠΑ ή το διεθνές πλαίσιο. Ε, υπάρχει ε, διαφάνεια με την οποία γίνονται διαπραγματεύσεις και χρησιμοποιείται η πυρονομοσύνη όλων των κρατών μελών. Και πολύ φυσικά συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Θα σας δώσω λοιπόν μια πρώτη εικόνα το πώς εφαρμόζεται στον προγραμματισμό αυτή η διαδικασία. Δηλαδή όταν πρόκειται να διαπραγματευτούμε τις ε, συμφωνίες τελικής σχέσης και γύρω στο Πάσχα του προσεχούς έτους θα σα ενημερώσουμε πιο λεπτομεριακά για το πώς λειτουργήσε κατά τη διάρκεια της ε, υλοποίησης. Πρόκειται λοιπόν για μια φωτογραφία κατά κάποιο τρόπο στο πρώτο στάδιο της όλης διαδικασίας ε, και θα δούμε πώς θα λειτουργήσει στο πλαίσιο αυτό, αλλά φυσικά θα γνωρίζουμε τις ε, εξελίξεις μακροπρόθεσμα. Υπάρχουν δύο βασικά στάδια. Το πρώτο ε, αφορά τέσσερις μελέτες που αξιολογούν το πρόγραμμα για την εφαρμογή του όλου μηχανισμού, το πλαίσιο λειτουργίας, τον κώδικα εφαρμογής και Νομίζω ότι αυτή η μελέτη έχει ήδη παρουσιαστεί σε εσά και αυτή η μελέτη που σας παρουσιάζω σήμερα είναι συνδεμένη με αυτήν και μας λέει τι, τι διδάγματα μπορούμε να συνάγουμε. Υπάρχουν φυσικά και άλλες μελέτες πιο πολιτικής ε, χρειάς. Τώρα, ο στόχος της μελέτης ήταν να αναπτύξει μια ανάλυση για το πώς ε, οι κανονιστικές ε, ρυθμίσεις και διατάξεις εφαρμόζονται στο πρόγραμμα περί αιρεσιμότητας. Ε, οι αιρεσιμότητες εξάντε, όπως εξήγησε ο καθηγητής, εμπλέκονται στην θέμα της περιφερειακής πολιτικής, αλλά υπάρχουν και άλλες μορφές ερεσιμότητας. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με ένα περιορισμένο εύρος τώρα ερεσιμότητας και θέλουμε να δούμε πώς αυτή η διαδικασία που ρυθμίζεται στο δικό μας επίπεδο μεταφέρεται, μεταφράζεται σε εθνικό και υποεθνικό υπερφυριακό επίπεδο. Ε, θα, δεν θα αναφερθώ στις ε, διαφορές που υπάρχουν ανάμεσα στα κράτη-μέλη και ε, το θέμα της ε, σχέσης ανάμεσα στα εταιρικέ συμφωνίες και το λειτουργικό πρόγραμμα, το επιχειρησιακό πρόγραμμα. Για να πετύχουμε αυτή τη μελέτη προσπαθήσαμε να εξετάσουμε όλες τις ε, εταιρικέ συμφωνίες και συμφωνίες συνεργασίας και πολύ διάφορα προγράμματα χρηματοδότησης Ένα σημαντικό στοιχείο που θα ήθελα να τονίσω είναι ότι η τελική μας έκθεση έγινε σε συνεργασία με τα κράτη-μέλη. Θέλαμε να έχουμε μια επιβεβαίωση των συμπερασμάτων μας. Η παρουσία που σας κάνω είναι πολύ συνοπτική, νομίζω ότι έχετε λάβει αντίγραφα. Είναι 150 σελίδες. Απλά θα σας αναφέρω κάποια από τα βασικά σημεία, τα σημεία κλειδί. Ε, είναι μια περίπου πλήρης εικόνα Φυσικά τα πράγματα δεν αλλάζουν αν λάβουν υπόψη όλα τα ολοκληρωμένα προγράμματα. Υπάρχουν πολλές μορφές ε, ρεσιμότητας, ε, όπως σας είπα. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, τις ιερεσιμότητες έχουν όμως ένα περιορισμένο στόχο και αυτός είναι να διασφαλίσουμε ότι οι προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση βρίσκονται στην θέση τους, είναι έτοιμες προκειμένου να μπορέσουμε να ε, χρηματοδοτούμε κάποια προγράμματα. Οι προϋποθέσεις λοιπόν υπάρχουν και άρα τα χρήματα θα δαπανηθούν με τρόπο σωστό. Αυτό βασίζεται φυσικά στην εμπειρία μας ε, εμπειρία μερικές φορές των Κομισιόν και των κρατών μελών και μερικές φορές πληροφορίες που έρχονται από τους ε, ενδιαφερόμενους. Και υπάρχουν δύο είδη. Υπάρχουν ε, θεματικές εξάντε αιρεσιμότητες που συνδέονται με ειδικέ μορφές χρηματοδότησης και υπάρχουν διαφορών ειδών. Τρεις-τέσσερις διαφορετικές μορφές στρατηγικής μορφής ε, όπου είδαμε στο παρελθόν την απουσία στρατηγικής από πλευράς πρωτών μελών όπου υπήρχαν ασυντόνιστες επενδύσεις ε, και το, το, των καινοτομίων είναι ένα άλλο παράδειγμα. Υπάρχουν ε, ερεσιμότητες όπου η υλοποίηση του ευρωπαϊκού κεκτημένου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την ουσιαστική δαπάνη των κονδυλίων οι οδηγίε ε, περί αποτελεσματικότητας, ε, τη της ε, ενέργειας είναι ένα παράδειγμα. Δεν θα το σε λεπτομέρειε. θέμα του περιβάλλοντος, το οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα. Εάν λοιπόν όλα αυτά δεν είναι έτοιμα από πλευρά κράτου μέλους, τότε δεν μπορούμε και να χρηματοδοτήσουμε. Υπάρχουν θεσμικές προποθέσει και όλοι θα σας πούν ότι οι θεσμοί είναι ένα θέμα κλειδί για την διασφάλιση αυτών των αυτής της αιρεσιμότητας. Τώρα στρατηγική, κανονισμοί, θεσμοί, όλα αυτά λοιπόν δεν έχει σημασία αν όλα βρίσκονται στα χαρτιά. Σημασία έχει να υπάρχει διοικητική ικανότητα για την ε, διαχείριση αυτών των ε, περιπτώσεων. Για μια ακόμα φορά αναφέραμε τις ε, εξάντε κονδυσιονάλες, εξάντε ερεσιμότητες, αλλά αυτές είναι προϋποθέσεις εξάντε όπως, όπως ανέφερα. Χρειάζονται κάποιες γενικές αρχές που θα πρέπει να εφαρμοστούν σε ό,τι αφορά τις ε, συγκεκριμένες ε, μορφές χρηματοδότησης τώρα. Εδώ είναι κάποια παραδείγματα για του είδους προϋποθέσεις θεωρούμε σημαντικές στον κανονισμό ε, στρατηγική μεταφορών, ε, περιβάλλον, ε, σύστημα δημοσίων προμηθειών, φιλικό προς την επιχειρηματικότητα, στρατηγικές για την καινοτομία κλπ. Αυτά είναι τα πρώτα στοιχεία που σας αναφέρω αναφορικά με τις ε, θεματικές αιρεσιμότητες και να ε, αναφερθώ τώρα στις γενικές ε, αιρεσιμότητες. Να πω ότι ένα από τα σημαντικά στοιχεία του κανονισμού δεν είναι μόνο η χρηματοδότηση, αλλά η χρηματοδότηση με κάποια συγκεκριμένη μορφή και σύμφωνα με τις αρχές Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν λοιπόν τρεις εξάντε αρεσιμότητες οριζόντιας φύσης ε, που είναι πολύ σημαντικές. Αυτό ε, ήταν αντικείμενο εκτενών συζητήσεων μεταξύ Συμβουλίου και Κοινοβουλίου και συνδέονται με την ικανότητα εφαρμογής ε, ε, θεματικότητας κατά των διακρίσεων και των και το θέμα είναι αν πρόκειται να επενδύσουμε σε ή οδήποτε τομέα θα πρέπει να τηρήσουμε αυτές τις αρχές και στο τέλος της διαπραγμάτευσης αυτά συμπεριλήφθησαν. Υπάρχουν και τρεις ακόμα, τρία ακόμα είδη εκ των προτέρων αρεσιμότητας που έχουν σημασία σχετικά με τα προβλήματα που είδαμε κατά την υλοποίηση των πολιτικών μας. Το είδαμε αυτό και με το ελεγκτικό συνέδριο σε, ε, σε περιπτώσεις ε, περιβάλλοντος, ε, κρατικών προμηθειών κλπ. Όλα σε αυτές λοιπόν εστίασαν στις διοικητικές ικανότητες. Δίνουμε έμφαση στην βελτίωση των αποδοτικότητας και εστιάσαμε ιδιαίτερα στην οριζόντια εξάντε αιρεσιμότητα και μιλάμε για δείκτες και στατιστικές. Τώρα, αυτή είναι η ιστορία της ε, εξάντε αιρεσιμότητας. Ε, το συγγνώμη, διότι η διαφάνεια δύσκολα είναι αναγνώσιμη. Βλέπουμε ότι μη πλήρωση των ε, αιρεσιμοτήτων εξάντε αφορούν τους τομείς ε, στατιστικών και δικτών και των δημοσίων προμηθειών. Βλέπουμε επίσης στο αριστερό τμήμα όπου υπάρχει το ζήτημα της ε, καταπολέμησης των διακρίσεων και των ε, αναπηριών βλέπουμε ε, περίπου 10 κράτη τα οποία δεν πληρούν ε, αυτά τα κριτήρια. Μία από τις σημαντικές πτυχές ε, της εξάντια είναι, να αποτελεί ένα είδος διάγνωσης, εργαλείου διάγνωσης. Ποιες είναι λοιπόν οι σημαντικές προϋποθέσεις για χρηματοδότηση. Σε καμία από τις οριζόντιες εξάντια δεν υπάρχει μόνο πράσινο. Άρα πολλά απομένουν να γίνουν. Εκ των προτέρων ε, χρησιμοποιείται για να δούμε πού βρίσκονται οι ελλείψεις ε, ε, για να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα του προγράμματος. Εδώ βλέπουμε μια ακόμα φορά την συχνότητα. <coughs> δεν θέλω να πω, μάλλον να πω κάτι τώρα σχετικά με αυτά που είπε ο κ. καθηγητής. Εδώ δεν ε, αντανακλάται η εφαρμοσιμότητα, αλλά η χρήση των διαφόρων μορφών χρηματοδότησης των προγραμμάτων. Όπως βλέπετε υπάρχουν πολλές θεματικές εξάντερεσιμότητες ε, για να φέρονται πηγές όπου έχουν ε, δαπανηθεί πολλά κονδύλια, όπου υπάρχει θεματική συγκέντρωση. Πρόκειται για περιοχές ε, που αφορούν την καινοτομία, ενέργεια, απόδοση της ενέργειας κλπ. Νομίζω ότι αυτός ο πίνακας ε, αντανακλά την κατανομή των πόρων. Μας λέει όμως ε, πολλά για το μέλλον, για το περαιτέρω προβληματισμό μας. Και αυτό νομίζω θα το δείξει ο επόμενο αγορητή. Εδώ είναι η ιστορία της εκπλήρωση. Ε, το ιστορικό μάλλον. Το πράσινο είναι εκπλήρωση, το κίτρινο είναι μερική και το κόκκινο δεν υπήρξε καμία εκπλήρωση των προσδοκομένων αποτελεσμάτων. Θα μπορούσα να πω πολλά πάνω στη διαφάνεια, αλλά θα θέλω να τονίσω πως ε, εάν πάτε κάτω, στο κάτω κομμάτι διαφάνειας, υπάρχουν περιοχές όπου λιγότερο από 20% και εδώ μιλάμε για προγράμματα <clears throat> για την, που, εκπληρούν, που πληρούν τις προϋποθέσεις της εξάντερης ημότητας, ε, το μέσο του ύδατος, ε, αλλά και τον ε, ενεργό γύρανση. Σε αυτές τις περιοχές λοιπόν σύμφωνα με τα κριτήρια που υιοθετήσαμε, που πρότεινε η Κομισιόν και συμφωνήσαμε με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπάρχουν σημαντικά προβλήματα και πολλά μπορούν να γίνουν. Αυτή είναι η τομή όπου το κίτρινο και το κόκκινο είναι προγράμματα δράσης προκειμένου να ε, διορθωθούν. Αυτή η ιδέα της εκ των προτέρων ερεσιμότητας είναι ένα εργαλείο διάγνωσης και θα πρέπει και μας δείχνει ότι πρέπει να αναλάβουμε δράση. Τα εντοπίζουμε στο τέλος, μάλλον στην αρχή του προγράμματος, συγγνώμη, ε, πριν ξεκινήσουμε την δαπάνη των κονδυλίων, προτού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα και εμπλακούν οι ελεγκτές για θέματα νομιμότητας και κανονικότητας. Αυτό ήταν το κομμάτι το περιγραφικό και για να ολοκληρώσω μερικά μηνύματα σχετικά με το κανονιστικό θέμα. που δεν βασίζεται μόνο στο τι μας λέει δεν είναι συμβουλές, αλλά τι μας λένε οι εμπλεκόμενοι στα προγράμματα αυτά της ρεσιμότητας αν είναι τα κράτη-μέλη, αν είναι οι υπάλληλοι της Κομισιόν. Ποια είναι τα μηνύματα λοιπόν. Πρώτο μήνυμα είναι ότι το των προτέρων είναι πολύ σημαντική για το πρόγραμμα και τη δαπάνη των πόρων. Ξέρουμε λοιπόν τι πάει καλά, τι πάει, δεν πάει καλά, αλλά θεωρείται μια πολύ σημαντική άσκησης, ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα. Το δεύτερο είναι μια διαδικασία εκμάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους. Δηλαδή είναι κάτι το νέο, αλλά προσφέρει και κάτι στον τρόπο με τον οποίο σκέφτονται την πολιτική. Ήταν ένα πρόγραμμα φιλόδοξο και πολλές προκλήσεις ε, για πολλά κράτη-μέλη προκειμένου να ελέγξουν αυτά τα θέματα και τις σχέσεις ανάμεσα στα διάφορα όργανα αλλά επίσης αποτελούσε πρόκληση για την Κομισιόν για τον τρόπο με τον οποίο θα έπρεπε να οργανωθεί και τον τρόπο με τον οποίο θα εργαστεί και συνεργαστεί με τα κράτη-μέλη. Νομίζω ότι αυτή είναι η πιο θετική πλευρά. Μιλάω για το φαινόμενο τη Κομισιόν. Σε πολλέ περιπτώσει αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ε, άλλοι λέμε επιδρά με το κράτο μέλο ε, θεωρείται μια διαδικασία σε βάθος ε, και το μήνυμα που λάβαμε πολλά κρατημέλη είναι ότι θα χρειαζόταν ίσως παρετέρω χρόνος ε, διάθεσή τους για να δουλέψουν πιο αποτελεσματικά, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα, χρειάστηκε να διαπραγματευτούμε τώρα πράγματα, ξέρουμε ποιες ήταν οι ε, καταστάσεις όπου τα, οι δέσμες και οι κανόνες εγκρίθηκαν κάπως γρήγορα έτσι έχουν τα πράγματα. Φυσικά θα μπορούσαν να έχουν γίνει καλύτερα, αλλά και αυτό φυσικά σε αυτό φυσικά βοήθησε η διαπραγμάτευση. Τώρα, τα δυνατά σημεία και οι αδυναμίες. Τώρα, σε αυτά τα δυνατά σημεία, αυτή εκ των προτέρων ερεσιμότητα συγκρινόμενη με προηγούμενες περιόδους υπάρχει ευρύτατη συνένεση ότι όλοι συνειδητοποίησαν πως το να δαπανίσουν, δαπανούν τα χρήματα σωστά δεν σημαίνει ότι απλά δαπανούνται. Θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προϋποθέσεις για να γίνει αυτή η σωστή δαπάνη, η κατάλληλη δαπάνη. Και να αντιμετωπίζουμε τα διάφορα προβλήματα γέρος. Ένα άλλο ισχυρό σημάδι είναι ότι οδηγεί στην ενισχυμένη συνεργασία ανάμεσα στα εθνικά και περιφερειακά επίπεδα. Τα τη μέλη αυτό δεν ήταν πάντα εύκολα, εύκολο να επιτευχθεί, αλλά όταν υπάρχει εθνική νομοθεσία και περιφερειακή δαπάνη, η τούμπαλη, οδήγησε όμως σε νέα μορφή αλληλεπίδρασης, και το είπα και προηγούμενα, άλλαξε τον τρόπο και το περιεχόμενο της συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης μεταξύ κράτη κρατών μελών και η Κομισιόν δεν ήταν πάντα εύκολο, αλλά εμπλούτησε την συζήτηση. Είναι σαφές ότι στη διαδικασία, το βλέπετε αυτό στη μελέτη, ότι στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης των προγραμμάτων και προσπαθούμε να πετύχουμε τις ε, εκ των προτέρων υπήρξε βελτίωση. Και αυτό έγινε αισθητό. Ειδικά είδαμε, προ, βελτιώσεις στην ε, πλήρωση των ε, προϋποθέσεων εξάντε, την χρηματοδότηση, αλλά και βελτίωσε την ε, θεσμικές και ικανότητες. Αν είχαμε έναν πίνακα επιτυχίας στην αρχή του προγράμματος και ένα στο τέλος, τότε θα βλέπαμε σημαντική βελτίωση μπορούσαμε να κάνουμε μια σύγκριση ενός τέτοιου πίνακα. Και τέλος, ε, τις ε, ελλείψεις ε, στα δυναμίες. Πρώτον, χρειάστηκε πολλούς πόρους από πλευράς κρατών μελών, ειδικά από τα κράτη-μέλη που επενδύουν. Αν πάμε στο θέμα της εξάντη και των πίνακα, η οι περισσότερες χώρες ε, ε, χρηματοδοτούν σε πολλούς τομείς. Και αυτό φυσικά ήταν ε, μια πρόκληση. Να πω ότι ήταν πολιτική πρόκληση, διότι μερικές φορές αφορούσε τομείς πολιτικά ευαίσθητους τα περισσότερα κράτη-μέλη. Να πω ότι θεωρήθηκε πως η πρόκληση και ο φόρτος εργασίας ήταν δυσανάλογος. Νομίζω ότι είναι νωρίς για να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτής της ε, εκ των προτέρων ρεσιμότητας, αλλά μπορούμε να δούμε γέρο πως ε, υπήρχαν θετικέ επιπτώσεις. Και αυτές οι θετικές επιπτώσεις ε, είχαν κάποιο κόστος και από πλευρά ε, κομισιών. Το μέλλον, το ερώτημα θα είναι πώς θα βελτιώσουμε αυτή την κατάσταση, αλλά στην επόμενη έκθεσή μας που θα φτάσει γύρω στον Μάρτιο-Απρίλιο θα ενημερωθείτε καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως είπατε, όσον αφορά τη διάγνωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δέχεται πια να δει τον ασθενή. Ο κύριος David Κόρνα τώρα, διευθυντής υπεύθυνο για την αξιολόγηση των συμφωνιών εταιρική σχέσης. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ε, ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε τη δυνατότητα που να ε, εκφράσω μια πρακτική ε, εμπειρία ε, στην Τσεχία. Θα παρουσιάσω, θα κάνω την παρουσίασή μου στα τσεχικά. Tak, děkuji za slovo ještě jednou. Budu pokračovat v českém jazyce. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να χρησιμοποιήσω την ε, μετρική μου γλώσσα για την παρουσίαση αυτή πριν σας δώσω συγκεκριμένες ε, πληροφορίες για τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες στη Δημοκρατία. Θα είναι χρήσιμο νομίζω να σας ε, αναφερθώ στις γενικές αρχές των εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων. Ο αρχικός στόχος των ερεσιμοτήτων αυτών ήταν η βελτίωση της ποιότητας των δημοσίων δαπανών, ειδικότερα στις περιόδους δημοσιονομικών ε, περιορισμών. Αυτό ήταν και σύμφωνο με τα αποτελέσματα, τα συμπεράσματα ε, που αφορούσε τον προπολογισμό του 2010, ένας από τους βασικούς στόχους που είναι πολύ σημαντικός για μας και που είναι και ε, ε πολύ ε, λογικός λόγω της συγκυρίας είναι η δυνατότητα άντλησης χρηματοδότησης μέσω των ερεσιμοτήτων αυτών, ώστε τα κονδύλια να χρησιμοποιούνται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και ο τρίτος στόχος ε, είναι το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες ε, υφιστάμενες υποχρεώσεις ε, σε κάποιους τομείς, ειδικότερα όσον αφορά την εφαρμογή της ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Σε μερικά κράτη-μέλη αυτή η νομοθεσία οι όροι της νομοθεσίας αυτής δεν έχουν ακόμη εφαρμοστεί και επίσης υπάρχει και η πέμπτη έκθεση συνοχής που καταδεικνύει ακριβώς αυτό το γεγονός. Θα ήθελα να σας δώσω λίγο περισσότερες πληροφορίες τώρα για τη συγκεκριμένη κατάσταση στην τσεχική δημοκρατία. Βλέπετε πώς έχουν τα πράγματα αυτή την εβδομάδα έχουμε τους 11 θεματικούς στόχους και βλέπουμε ότι σχεδόν όλοι ε, οι όροι έχουν ε, ε, ε, γίνει σεβαστή 40 όροι και μόνο 8 στόχοι δεν έχουν ε, εκπληρωθεί, 8 ε, όροι δεν, έχουν, δεν πληρούνται ακόμη. Και υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι αυτή τη στιγμή την κάνουν επαλήθευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τρεις θεματικοί όροι που δεν έχουν πληρωθεί. Νομίζω λοιπόν ότι πρόκειται για μία επιτυχημένη ιστορία. Είπα ότι υπάρχουν μόνο τρεις στόχοι που εν μέρη έχουν πληρωθεί είναι οι δημόσιες μεταφορές, η δημόσια διακυβέρνηση και οι δημόσιες προμήθειες. Και πιστεύουμε ότι μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους θα έχουν εκπληρωθεί ε, και αυτοί οι όροι ε, πλήρως. Ε, υπάρχουν και κάποιες επαληθεύσεις που γίνονται αυτή τη στιγμή όσον αφορά τη διαχείριση των υδάτων, το, τις σιδηροδρομικές μεταφορές ή ο τομέας της υγείας, μεταξύ άλλων, που αυτή τη στιγμή βρίσκονται υπό επαλήθευση. Αυτά ήταν ορισμένα αριθμητικά στοιχεία από τις στατιστικές μας. Θα ήθελα να σας πω όμως ε, ορισμένα πράγματα και για το σύστημα το οποίο ε, χρησιμοποιούμε από το 2011. Το πρώτο ε, σημαντικό είναι να ε, εντοπίσουμε τους αρμόδιους φορείς ε, στην Τσεχική Δημοκρατία. Το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι ο βασικός φορέας, είναι ένας ε, φορέας γενικός που είναι επικεφαλής αυτών των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων και υπάρχουν κάποιοι επιμέρους αρμόδιοι φορείς που είναι υπεύθυνοι για την εκπλήρωση των όρων αυτών. Επίσης υπάρχει και ε, το επίπεδο της υποστήριξης των άλλων εμπλεκομένων φορέων. Υπάρχουν και άλλοι φορείς λοιπόν που είναι σημαντικοί για την εκπλήρωση των ε, όρων και προϋποθέσεων και πρέπει να λάβουμε υπόψη το γεγονός ότι οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες υπερβαίνουν τη δομή εφαρμογής ε, κατά το μεγάλο ποσοστό τους. Δηλαδή μερικές φορές είναι πάρα πολύ δύσκολο όλες αυτές οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες να τις καλύψουμε γιατί πρέπει κανείς ε, να προσκαλέσει σε ένα τραπέζι ε, πολλούς φορείς οι οποίοι πρέπει να συντονιστούν, να συνεργαστούν και να ορίσουν μια κοινή στρατηγική. Επίσης, πολλές φορές υπάρχει ένα πρόβλημα ε, ευθύνης. Αν υπάρξει κάποιο, κάποια αναστολή ε, πληρωμής, για παράδειγμα, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Εδώ βλέπετε έναν πίνακα για τον τρόπο με τον οποίο συμμετέχουν στη διαδικασία οι αρμόδιοι ε, φορείς. Βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά ακρονίμια. Θα ήθελα να σας δείξω ότι είναι μεγάλος ο αριθμός των ε, φορέων που θεωρούνται υπεύθυνοι για τη διαδικασία αυτής της δεχική δημοκρατία. Βλέπετε λοιπόν ε, ότι είναι οι αρμόδιοι φορείς, ε, συνεργαζόμενοι φορείς και αυτοί οι δύο πίνακες που σας δείχνουμε είναι γενική, αλλά μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα. Το Υπουργείο Εμπορίου και Βιομηχανίας ή το Υπουργείο Κοινωνικών Υποθέσεων, αυτά τα Υπουργεία είναι υπεύθυνα για κάποιες ε, αιρεσιμότητες. Ε, το ίδιο ισχύει για το Υπουργείο Γεωργίας που είναι υπεύθυνο για κάποιες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Ε, συνολικά υπάρχουν 11 υπουργεία και υπάρχει επίσης και το γραφείο της κυβέρνησης. Όλα τα Υπουργεία συμμετέχουν λοιπόν στη διαδικασία. Αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με το, τη Στατιστική Υπηρεσία της Τσεχίας και το Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Τσεχίας και συνεργαζόμαστε και με περιφερειακούς εταίρους. Το σύστημα είναι πολύ ε, σταθερό, η συμμετοχή των εταίρων είναι πολύ μεγάλη. Μερικές φορές αυτό σημαίνει βέβαια ότι υπάρχουν και πολύ δύσκολες διαπραγματεύσεις. θα ήθελα τώρα να σας δείξω κάποιες πλατφόρμες και κάποιες δομές σημαντικές που πρέπει οπωσδήποτε να συμπεριληφθούν στη διαδικασία. Κάποιες από αυτές είναι πολύ σημαντικές για τις διαδικασίες ε, αδειοδότησης και μερικές φορές ε, ήρθαμε σε διαβούλευση με τους φορείς αυτούς. Βλέπετε το κατάλογο των ε, ε, φορέων αυτών, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παράδειγμα, υπάρχει ε, η κυβέρνηση της Αιχικής Δημοκρατίας και άλλοι φορείς. Να σας εξηγήσω τώρα με απλό τρόπο το σύστημά μας. έχουμε προετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης, το οποίο εγκρίθηκε από την κυβέρνηση και αυτό το σχέδιο δράσης Είναι το σημείο αφετηρίας ε, για τη δουλειά μας. Το σχέδιο δράσης στη συνέχεια εξελίσσεται σε σχέση με τις εξελίξεις στις διάφορες τομεϊκές πολιτικές και επίσης και σε σχέση με την εξέλιξη των εκτοπροτέρων αιρεσιμοτήτων, κάποιο, ένα μέσο που είναι πολύ σημαντικό για την τσεχική δημοκρατία και όχι μόνο στον τομέα αυτό είναι το ενσωματωμένο σύστημα διαχείρισης κινδύνου, το οποίο είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα για τα επιχειρησιακά προγράμματα. Ε, πρόκειται για την αξιολόγηση κινδύνων ε, σε οριζόντιο επίπεδο. Ε, το συμβουλευόμαστε συχνά, όπως επίσης και το πρόγραμμα διαχείρισης κινδύνου ε, που εξετάζεται ε, και από την ε, κυβέρνηση. Το σύστημα λοιπόν αναφέρεται σε κινδύνους όπως επίσης και σε προτάσεις αντιμετώπισης των κινδύνων αυτών. Υπάρχουν και κάποια χρονοδιαγράμματα. Εν ολίγης δηλαδή, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, τι μέσα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το κάθε πρόβλημα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το μέσο για μας. Όσον αφορά την παρακολούθηση τώρα. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Είναι πολύ σημαντικό και για τους υπεύθυνους ε, φορείς. Εμείς αποφασίσαμε στη Τσεχική Δημοκρατία να καταρτίζουμε μία τριμηνιαία έκθεση παρακολούθησης, ε, συμπεριλαμβάνει πληροφορίες ε, για την ε, τρέχουσα κατάσταση, για τις συζητήσεις μεταξύ των φορέων, επίσης εντοπίζει προβλήματα και πιθανές λύσεις. Και πλησιάζουμε τώρα και στο προ... στην προθεσμία μας που είναι το τέλος του 2016. Γι' αυτό ετοιμάζουμε τώρα και μία ειδική έκθεση κάθε μήνα. Και υποβάλλουμε αυτή την έκθεση κάθε μήνα στην Τσεχική Δημοκρατία. Θα ήθελα επίσης να σας αναφερθώ στις τριμερείς συζητήσεις που είναι πάρα πολύ σημαντικές ώστε οι οικονομικοί και κοινωνικοί μας εταίροι που μπορούν επίσης να παρέμβουν σε ειδικού ε, τομείς ε, είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό. Πλησιάζω στο τέλος της παρουσίασής μου. Θα ήθελα να ολοκληρώσω αναφερόμενος ε, στα ισχυρά αλλά και στα ε, αδύναμα σημεία της στρατηγικής μας, μπορούμε να δούμε πολλά ωφέλη. Θα σας δώσω και κάποια παραδείγματα μετέπειτα. Ένα από τα ωφέλη είναι ότι η στρατηγική προσέγγιση και προγραμματισμός ενισχύονται πριν από την αρχή των ε, projects. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι υπάρχει θετική πίεση για την εφαρμογή αυτών των στρατηγικών, την εφαρμογή τους στην πράξη, η τσεχική δημοκρατία έχει εκπονήσει 35 έγγραφα στρατηγικής και είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι δεν έχουμε προγράμματα περιφερειακής συνεργασίας, ε, έχουμε θεματικά προγράμματα συνεργασίας και η στρατηγική καταρτίζεται μόνο σε εθνικό επίπεδο. Οπότε το στρατηγικό επίπεδο είναι πολύ σημαντικό και το άλλο επίπεδο είναι το επίπεδο της νομοθεσίας. Σε μερικές περιπτώσεις οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ε, πίεσαν για αλλαγές στο νομοθετικό μας σύστημα και υπάρχει επίσης και η μεταγραφής της ενωσιακής νομοθεσίας ή προετοιμασίας ειδική νομοθεσίας στην Τσεχική Δημοκρατία, για παράδειγμα, τροποποίησε 10 νόμους για να μπορέσει να ε, εφαρμόσει τις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες υπάρχει και κάποια προστιθέμενη αξία σε αυτό και θα ήθελα να αναφερθώ ε, σε αυτό που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως ότι υπάρχουν κάποιες ε, καινοτομίες όπως για παράδειγμα ε, ε τις, οι αρχές της εφιούς εξειδίκευσης. Εμείς θέλουμε να εμπλέξουμε και συνεργάτες από το περιφερειακό επίπεδο ήταν απαραίτητο να ευθυγραμμίσουμε την ε, περιφερειακή μεθοδολογία με την ε, εθνική μεθοδολογία, αλλά επειδή το ε, σύστημα ήταν τόσο περίπλοκο, είναι δύσκολο να αξιολογηθεί το σύστημα στο σύνολό του αυτή τη στιγμή. Επίσης πρέπει να πούμε ότι η αποτελεσματικότητα της διοίκησης έχει αυξηθεί. Για παράδειγμα, οι δημόσιες προμήθειες, οι, ε, στους τομείς της ε, αναπηρίας, ε, της ε, διάκρισης μεταξύ των φύλων, ε, μπορέσαμε λόγω αυτών των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων να αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα. Επίσης υπήρξε μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των εμπλεκομένων φορέων εντός ε, της δομής εφαρμογής και μπορούμε να δούμε ότι σε μερικές περιπτώσεις η πολιτική συνοχής ε, προσπαθεί να μην είναι ε, τόσο περιοριστική, προσπαθεί να συμπεριλάβει πολλούς εταίρους και αυτό νομίζουμε ότι είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν συζητούσαμε συνεδριάσεις μας τις αιρεσιμότητες αυτές δεν μιλούσαμε μόνο για προβλήματα, μιλούσαμε και για τα σχετικά ε, ζητήματα και αυτό είναι ένας πολύ καλός τρόπος ε, να προχωρήσουμε. Γι' αυτό θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ισχυρό σημείο του συστήματός μας. Υπάρχουν επίσης νέα σημεία ε, επαφών που ήταν υπεύθυνα για τα θέματα ισότητας των φύλων, για παράδειγμα. Υπάρχουν νέα λοιπόν σημεία ε, επαφών, contact points, τα οποία ήταν υπεύθυνα για την παρακολούθηση των ε, ε, ε, της ισότητας των φύλων και γι' αυτό, γι αυτό πιστεύουμε ότι είναι ένα καλό παράδειγμα. Θα ήθελα να αναβρεθώ τώρα ε, και σε ορισμένους περιορισμούς, ή πιο αδύναμα σημεία του συστήματός μας. Καταρχάς, κάποια προβλήματα δημιουργούνται λόγω ε, αιρεσιμοτήτων σε εθνικό επίπεδο. Το εθνικό επίπεδο λοιπόν είναι υπεύθυνο για την επίλυση του προβλήματος αυτού. Όμως, σε μερικές περιπτώσεις, οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες έχουν κάποιους περιορισμούς. Θα προσπαθήσω να σας δώσω παραδείγματα. Μερικές φορές το πρόβλημα είναι έλλειψη προβλεψιμότητας όλων των προϋποθέσεων. Μερικές φορές ε, άλλαξαν ε, οι προϋποθέσεις κατά τη διάρκεια του έργου. Ξεκινούμε, ε, ξεκινήσαμε το 2012 με τις εκνοπροτέρων ερεσιμότητες, κάναμε κάποιες προετοιμασίες, όμως μετά έπρεπε να κάνουμε προσαρμογές και να κάνουμε κάποιες αλλαγές. Κάποιο ακόμη ισχυρό μας σημείο, ε, συγγνώμη, αδύναμό μας σημείο, αδύνατο μας σημείο είναι το υπερβολικό διοικητικό άχθος. Αυτό έχει κάποια προστιθέμενη αξία, αλλά δημιουργεί και προβλήματα. Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα του διοικητικού άχθους. Πρέπει να μάθουμε πώς θα διαχειριζόμαστε τις διοικητικές απαιτήσεις. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι μερικές φορές η δυνατότητα απορρόφησης όλων των ε, προϋποθέσεων και προσαρμογής της νομοθεσίας σε περιορισμένο χρονικό διάστημα. Ε, υπάρχουν ε, και άλλα ε, προβλήματα σε επιχειρησιακό επίπεδο και νομίζουμε ότι πρέπει να συζητηθούν αυτά τα θέματα στο μέλλον, να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, για παράδειγμα διαφορετικές προσεγγίσεις ε, στις υπηρεσίες, να έχουμε μια μεγαλύτερη εμβέλεια απαιτήσεων, μερικές φορές παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτό. Μερικές φορές ε, παίρνει ένα μήνα, άλλες φορές ένα χρόνο. Ένα ακόμη πρόβλημα είναι ο ορισμός νέων απαιτήσεων. Για παράδειγμα, υπήρχε ένας στόχος ε, για την συμπερίληψη των Ρωμά. Μας ζητήθηκε να προετοιμάσουμε μία νέα στρατηγική, αλλά μας ζητήθηκε να ε, δημιουργήσουμε και ένα νέο σύστημα παρακολούθησης με πάρα πολύ λεπτομερείς προϋποθέσεις, ειδικού δείκτες, για αυτά, αυτό το συγκεκριμένο στόχο. Επομένως, μερικές φορές είναι πολύ λεπτομερές θα ήθελα λοιπόν να σας πω και κάποιες προτάσεις μας για το μέλλον. Θεωρούμε ότι το σύστημα είναι θετικό, αλλά πιστεύουμε ότι για το μέλλον αναγκαίο είναι να έχουμε κάποιες δικλείδες ασφαλείας ώστε να δουλεύουν τα πάντα σωστά. Απλοποίηση. Για παράδειγμα, θα ήταν καλύτερα εάν ο αριθμός των εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων μειωθεί αν όμως είναι και καλύτερα ορισμένες ε, οι, προϋπο- οι αιρεσιμότητες αυτές από την αρχή, θα ήταν καλύτερα. Μικρότερος αριθμός λοιπόν εκ των προτέρων αιρεσιμοτήτων, οι οποίες θα ορίζονται και με καλύτερο τρόπο από την αρχή, με, με σαφέστερο τρόπο. Δεύτερος τομέας είναι η προβλεψιμότητα. Η διαδικασία πρέπει να είναι προβλέψιμη. Μερικές φορές αλλάζουν οι κανόνες κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Και μερικές φορές είναι σημαντικό να ε, γίνονται σεβαστές και οι απόψεις των κρατών μελών. Ε, η ομοιογένεια, μια κάπως πιο συνεπής προσέγγιση, αλλά πρέπει να λαμβάνετε υπόψη ότι και κάθε χώρα είναι διαφορετική. Μερικές φορές δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε μια ε, προσέγγιση που να ταιριάζει σε όλους. Νομίζω ότι και κάποιος προλαλής σας συνάδελφος ε, ανέφερε ότι είναι ε, υπάρχουν ε, ιδιαιτερότητες στις διάφορες χώρες και ότι χρειάζεται μια πιο ε, προσαρμοσμένη προσέγγιση. Η εμπιστοσύνη και η εκμάθηση επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικά. Πιστεύουμε ότι εκ των περαιτέρων αιρεσιμότητες είναι σημαντικές είναι, ότι, είναι γεγονός ότι βελτιώνουν την εμπιστοσύνη και την εκμάθηση. Θεωρούμε επίσης ότι δεν θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ε, μόνο ως κυρώσεις. Ε, νομίζουμε ότι θα έπρεπε μάλλον ε, να ενισχύσουμε το περιβάλλον στο οποίο υφίστανται, να είναι πιο έντονες οι αλλαγές. Θα πρέπει δηλαδή να είναι κάτι θετικό και όχι μόνο κυρώς. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Με χαρά θα απαντήσω σε ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτές τις λεπτομερέστατες παρουσιάσεις. Τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη της Επιτροπής μας. Έχω ήδη τον κατάλογο των ε, μέλων που επιθυμούν να μιλήσουν. Ο κύριος Όλμπριχτ έχει το λόγο. Παρακαλώ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Καταλαβαίνω πως εκ των ε, προτέρων αιρεσιμότητα είναι η άλλη όψη του νομίσματος της ε, ε, περιφερειακή πολιτικής. Μιλάμε για την πολιτική του Ρωμά κτλ. Το πραγματικό ερώτημα όμως εδώ νομίζω είναι το ποια είναι η σχέση ανάμεσα ε, στα, στις εκ των προτέρων αιρεσιμότητες και τα αποτελέσματα. Όταν δηλαδή πληρούνται οι προϋποθέσεις, τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Από τα διαρθρωτικά ταμεία ήδη μας ήταν γνωστό αυτό. Απλά πήρε άλλο όνομα και το σύστημα είναι λίγο διαφορετικό. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω τους ομιλητέ το εξή. Έχουμε κάποιες αποδείξεις για το ότι πληρούνται οι για το ότι όταν πληρούνται οι προϋποθέσεις τα αποτελέσματα είναι καλύτερα. Εάν ισχύει αυτό, τι είναι πραγματικά ε, η εκ των προτέρων αρεσιμότητα. Είναι κάποιες κατευθυντήριες γραμμές, είναι κάποιες απαιτήσει. Δηλαδή, ε, θέτουμε κάποιες προϋποθέσεις, εφόσον αυτές πληρούνται μπορούμε να αρχίσουμε ή ε, μιλάμε στο στάδιο της εφαρμογής. Το εξάντε εκ των προτέρων σημαίνει ότι πληρείται η προϋπόθεση, αλλά εάν αλλάξουν οι συνθήκες στην πορεία, αυτό έχει τελειώσει. Δεν μπορείς να αλλάξεις κάτι εκ των προτέρων. Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα εδώ, μπλέκονται τα πράγματα, ε, πάβει να είναι ε, εκ των προτέρων αιρεσιμότητα όταν αλλάζει την πορεία. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θέλω να ρωτήσω πόσο καιρό χρειάζεται μέχρι να φτάσουμε σε ένα στάδιο που θα πληρούνται όλες οι προϋποθέσεις για να περάσουμε στην συνέχεια. η εκ των προτέρων αρεσιμότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τα συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά ε, και με πολλά περισσότερα. Δεν μπορούμε, για παράδειγμα, ε, να μετρήσουμε ποσοτικά την διοικητική ικανότητα. Μπορούμε φυσικά να αρχίσουμε μια συζήτηση, όμως πρέπει να έχουμε υπόψη μας και το ότι υπάρχει ενδεχομένο αλλαγών. Και επίσης να ρωτήσω και το άλλο. Ποιο είναι ο ρόλο τη εκ των προτέρων αιρεσιμότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλαδή θέτει κάποιες προϋποθέσεις για να χρηματοδοτήσει ε, προγράμματα. Τα χρήματα αυτά όμως προέρχονται από τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις δεν παίρνεις χρήματα, δικά μας χρήματα. Ε, ευρωπαϊκά. Υπάρχει μια διαφορά όταν αρχίζει κάτι από τη βάση προς τα πάνω. Πρέπει, όπως είπατε και στην παρουσίασή σας, να είναι προσαρμοσμένες οι προϋποθέσεις της ανάγκης. Μετά, είναι υποχρεωτικός ο χαρακτήρας τους ή είναι απλά έτσι, μία σύσταση, κατευθυντήριες γραμμές πρέπει όλες οι προϋποθέσεις να πληρούνται ή ορισμένες από αυτές. Πρέπει λοιπόν να έχουμε απάντηση σε αυτό το ερώτημα, διότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά, θεσμικά οργανά, το Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατηγορούνται για την ε, κακή χρήση των ε, διαρθρωτικών ταμείων εξαιτία αυτής της εκ των προτέρων αρισιμότητας. Και γίνεται λόγος για ε, υλοποίηση κατά τη διάρκεια και όχι πριν. Είναι λοιπόν ένα πολύ περίπλοκο ζήτημα, το οποίο πιστεύω θα έπρεπε να είχαμε εξετάσει πολύ νωρίτερα, να είχε γίνει κατάλληλη συζήτηση με τα κράτη-μέλη, προτού οδηγηθούμε στην πολιτική απόφαση για τις ε, κατευθυντήριες γραμμές. Και πιστεύω πως ε, όλοι οι ομιλητές είχαν πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, διότι πραγματικά ε, εάν δεν υπήρχε η περιφερειακή πολιτική θα είχαμε σοβαρό πρόβλημα. Βρισκόμαστε σε πολύ δύσκολη θέση και νομίζω πως ε, είναι ό,τι χειρότερο να περιπλέξουμε τα πράγματα ακόμα περισσότερο. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Μαλέτης, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις τους. Συμφωνώ και εγώ με τον ε, κύριο Όλμπριχτ. Έχουν μειωθεί εκ των προτεραιών αρισιμότητες για τον επόμενο ε, ορίζοντα. Τώρα βρισκόμαστε στο στάδιο της ενδιάμεσης αναθεώρησης. Το 2017 θα έρθει και πρέπει να δούμε αν αυτές οι ε, προϋποθέσεις πληρούνται σε πολλές θεματικές προτεραιότητες. Αλλά νομίζω πως ε, πρέπει να υιοθετήσουμε μια πιο διαφορετική προσέγγιση σε σχέση με τις προτεραιότητες. Υπάρχουν οι προτεραιότητες που έχουν πολύ μεγάλη συχνότητα, το 1,1 ας πούμε έρευνα και ανάπτυξη, καινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ε, ψηφιακή ανάπτυξη, ενεργειακά ζητήματα. Αυτές εκπροσωπούνται ε, αρκετά. Όμως αν δούμε και τον άλλο πίνακα που παρουσιάσατε, βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλές εκ των προτέρων αρισιμότητες που δεν πληρούνται. Ακόμα δηλαδή δεν υπάρχει υλοποίηση. Και θα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, μία μέθοδο υλοποίησης παράλληλα με την ε, προσπάθεια να τηρήσουμε τις άλλες προϋποθέσεις. Ε, τώρα υπάρχουν και κάποιες άλλες θεματικές προτεραιότητες, λιγότερο σημαντικές, για τις οποίες ήδη πληρούνται κάποιες ε, προϋποθέσεις από αυτές τις ε, εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Πώς μπορούμε λοιπόν να συντονίσουμε όλα αυτά, να γίνει μια εναρμόνιση έτσι ώστε να αποφύγουμε το πρόβλημα της απορρόφησης και της υλοποίησης. Χρειάζεται να βρεθεί μια ισορροπία ανάμεσα στην έγκαιρη υλοποίηση και την κατάλληλη υλοποίηση. Και πρέπει να σκεφτούμε πέρα από τον ε, χρονικό ορίζοντα του 2020, διότι αν αλλάξουν οι προϋποθέσεις για την επόμενη προγραμματική περίοδο θα έχουμε πάλι τα ίδια προβλήματα. Πρέπει να δούμε λοιπόν τι θα κάνουμε, αν θα συνεχίσουμε όπως τώρα ή αν θα ζητήσουμε από τις χώρες να δημιουργήσουν νέες στρατηγικές για τους ίδιους τομείς. Αν θα πρέπει να τους ζητήσουμε να αρχίσουν από την αρχή την κατάρτιση νέων εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων για την επόμενη περίοδο. Είναι πολύ δύσκολη, περίπλοκη πολιτική και κάθε φορά παρατηρούνται αυτές οι καθυστερήσεις στην υλοποίηση και στην απορρόφηση. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Νίλσεν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω πως δεν υπάρχει σου ειδική διερμηνία, θα προσπαθήσω λοιπόν να μιλήσω αγγλικά. Και εγώ συμφωνώ με τον Γιάνν Όλμπριχτ. Είναι εξαιρετικά σημαντική αυτή η συζήτηση για την επόμενη περίοδο της πολιτικής συνοχής. Και υπάρχουν προβλήματα που χρειάζονται επίλυση. Δύο θέματα θέλω να αναφέρω τα οποία έχουν κάποια έμεση σχέση. Καταρχάς, για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα ήθελα να πω ότι πριν από δύο εβδομάδες συναντήθηκα με την κυρία Όλσον, την σύμβουλο του κυρίου Γιούνκερ στον κοινωνικό πυλώνα και μου είπε ότι ό,τι και αν κάνουμε πρέπει να θεωρούμε την κοινωνική πολιτική ε, παραγωγική για την οικονομική ανάπτυξη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Άνοιξη είπε το ίδιο, ότι χρειάζεται η πολιτική συνοχή, χρειάζεται γιατί επηρεάζει τις εξελίξεις. Φυσικά και δεν είναι καινούριο αυτό, διότι ήδη από τη δεκαετία του 90 είχαμε τονίσει τη σημασία ε, των, κοινωνικών, ε, των Ταμείων Κοινωνικών Επενδύσεων το πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε διάφορους, ε, διάφορες ομάδες όπως ανέργους για παράδειγμα για να τους ξαναβάλουμε στην ε, αγορά εργασία. Γι' αυτό λοιπόν δεν είναι αλήθεια ότι η κοινωνική πολιτική αποτελεί παραγωγικό παράγοντα, επηρεάζει την πολιτική συνοχής. Έπειτα να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Νομίζω καταρχάς πως όλοι συμφωνούμε πως η ε, η ικανότητα των ε, περιφερειών έχει πολύ σημαντικό ρόλο. Εάν θέλουμε επιτυχημένη πολιτική, πρέπει να δούμε και την διοικητική ικανότητα στις περιφέρειες. Δεν θα έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε τα προγράμματα τεχνικής υποστήριξης και στις περιφέρειες. Διότι έχω την εντύπωση ότι τα κράτη-μέλη χρησιμοποιούν αυτήν την τεχνική στήριξη για να χρηματοδοτήσουν τις διαφορές ε, εθνικές υπηρεσίες και όχι για να αυξήσουν τις ε, δυνατότητες των περιφερειών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βανίστελ Ρόι. Ευχαριστώ πολύ που ήρθατε σήμερα και μας δώσατε τη δυνατότητα να σας ακούσουμε. Είμαστε σε μια εποχή που πολλές φορές χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε το ένστικτό μας ε, στη χάραξη πολιτικής. Και νομίζω πως εδώ φαίνεται πως η μέθοδος που χρησιμοποιούμε είναι μεν πολύπλοκη, όμως τα αποτελέσματά της είναι θετικά. Ακόμα είναι βέβαια λίγο βέβαια τα πράγματα, είναι σαν ένα μαύρο κουτί που δεν έχουμε ανοίξει Όμως χρειάζεται να υπάρχουν ισχυρές συμμαχίες και συμφωνίες για να έχουμε αποτελέσματα. Βλέπω ότι γίνεται κατά τη διάρκεια της Σλοβακικής Προεδρίας, το Συμβούλιο και βλέπω ότι υπογραμμίζουν, τονίζουν αυτήν την προσέγγιση με τις ε, εκ των ε, προτέρων αρισιμότητες. Και άκουσα και τον ε, Τσέχο συνάδελφο, λέει τα ίδια. Υπάρχει προστιθέμενη αξία. Αυτό είναι θετικό νομίζω, τουλάχιστον αυτήν την εντύπωση έχω και όταν αργότερα θα ψηφίσουμε την έκθεση για την κατάσταση των επιχειρησιακών προγραμμάτων, για τα νέα προγράμματα τεχνικής ε, υποστήριξης και για την απορρόφηση. Ε, νομίζω λοιπόν ότι πρέπει να καταφέρουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο γι' αυτό, διότι δεν μπορούμε να περιμένουμε. Δεν έχουμε το χρονικό περιθώριο να περιμένουμε 7 χρόνια, 6 χρόνια. Όχι, αυτή τη στιγμή θέλουμε άμεσες λύσεις και οι πολιτικοί πρέπει να δρουν άμεσα και όχι να ε, χρονοτριβούν σχεδιάζοντας πολιτικές. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω και εγώ τους ομιλητές ε, τα εξής. Πώς μπορούμε αυτά τα θετικά ωφέλη να τα δρομολογήσουμε ταχύτερα. Πώς ε, γίνεται να το κάνουμε αυτό. Το 2017, όπως ξέρετε, θα είναι ένα έτος με νέες προτάσεις, με τις ε, νέες προτάσεις για την πολιτική συνοχής, για το φόρουμ συνοχής. εδώ βλέπουμε ότι μας λέτε πως μετά την ανάλυση βλέπουμε υπερβολική γραφειοκρατία, αυξημένο διοικητικό άχθος, ότι δεν δίδονται προτεραιότητες ε, όπως ε, θα έπρεπε κτλ. κτλ. Βλέπουμε λοιπόν αυτά τα λόγια, αυτά τα συμπεράσματα, αλλά θα μπορούσαμε επιτέλους να περάσουμε από την θεωρία στην πράξη. Γιατί το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων είναι έτσι κάπως γενικό, δεν ε, μπορούμε να το συσχετίσουμε με συγκεκριμένα προγράμματα, συγκεκριμένα έργα, συγκεκριμένους εταίρους, είναι έτσι γενικό και αόριστο. Για να χαϊδεύει τα αυτιά μας δηλαδή. Ε, πρέπει να περάσουμε επιτέλους από τις εκ των προτέρων αρισιμότητες τα αποτελέσματα και να επιταχύνουμε. Θα μπορούμε να επιταχύνουμε εγκαίρως, διότι εγώ βλέπω βέβαια τα ε, μικρά δομικά στοιχεία. Βλέπω τα τουβλάκια, δεν βλέπω το σπίτι. Αυτό λοιπόν είναι το κύριο ερώτημα που θέλω να σας θέσω. Ε, κύριε καθηγητά Σπάν, μας είπατε για τις Ηνωμένε Πολιτείες και το παράδειγμα εκεί. Υπάρχει κάποιο σύστημα, κάποια μέθοδος ε, που μπορούμε και εμείς να υιοθετήσουμε ως προς την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτσι ώστε να επιταχύνουμε τα αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να περιμένουμε να έρθει το 2020 και μετά να αρχίσουμε να λέμε ναι υπάρχουν 21 δις αποθεματικό και μπορούμε να κάνουμε αυτό και εκείνο. Όχι τότε θα έχουμε ένα νέο κοινοβούλιο. Το 2019 έχουμε ευρωεκλογέ. Σας παρακαλώ λοιπόν τα αποτελέσματα να είναι πιο συγκεκριμένα, να έρθουν συντομότερα, να αρχίσουμε ήδη τη συζήτηση στις αρχές του νέου έτους. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ευχαριστώ πολύ κύριο Σέτμαν. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τους ομιλητές για την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Σίγουρα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εκ των προτέρων αρισιμότητα είναι αναγκαία για να εφαρμόσουμε τις πολιτικές που συζητούμε εδώ. Ε, φυσικά και καταλαβαίνω και συμφωνώ με τον κύριο Όλμπριχτ και με τους άλλους συναδέλφους ευρωβουλευτές, αλλά δεν νομίζετε πως αυτή η μορφή της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περιφερειακή πολιτική στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα οδηγήσει στην επιβολή κάποιων ε, κατηγοριών που θα χρησιμοποιηθούν από τις ε, εθνικές κυβερνήσεις για τις περιφέρειες. Δεν θα οδηγήσει δηλαδή αυτό σε προβλήματα στο ότι οι περιφέρειες δηλαδή, οι διάφορες χώρες θα αρχίσουν να καταρτίζουν τις στρατηγικές τους με βάση αυτές τις εκ των προτέρων αρεσιμότητες και όχι με βάση τις πραγματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφέρειες. Δεν θα οδηγηθούμε δηλαδή στην απαλυφή της διαφορετικότητας, της πολυμορφίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πολλές φορές αυτό βλέπουμε να συμβαίνει, ότι δύο περιφέρειες που διαφέρουν κατά πολύ, όταν έχουν μια εκ των προτέρων αιρεσιμότητα, αρχίζουν να καταρτίζουν προγράμματα, να σχεδιάζουν πολιτικές, τα οποία δεν είναι προσαρμοσμένα στις πραγματικές τους ανάγκες, αλλά ε, στις προϋποθέσεις. Και νομίζω ότι ο καθηγητής ε, Σπάν μας είπε ότι στις ΗΠΑ είναι προσανατολισμένοι στο αποτέλεσμα και όχι στην ε, αξιολόγηση του κατά πόσο πληρούνται εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Εγώ πιστεύω πως αυτή είναι η σωστή προσέγγιση. οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες, έτσι όπως είναι τώρα, θα οδηγήσουν στην απώλεια της ε, πολυμορφίας. Και όταν αρχίσουμε να εφαρμόζουμε προγράμματα τέτοιου τύπου στις ε, διάφορες περιφέρειες, θα, θα δολοφονήσουμε αυτόν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα. Δεν θα υπάρχει πλέον ευελιξία στη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων όταν είμαστε δεμένοι χειροπόδαρα σε αυτές τις εκ των προτέρων αρεσιμότητες. Υπάρχουν ε, δεδομένα που αλλάζουν κατά τη διάρκεια μιας επταετούς περίοδου Και μπορεί καμιά φορά η αξιολόγηση να είναι αρνητική ή έστω να μην είναι θετική. Η αξιολόγηση εννοώ των προγραμμάτων που υλοποιούνται. Αλλά όπως και να έχει, σα ευχαριστώ για τις ε, πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Βόν έχει το λόγο τελευταίος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς ε, άργησα. Είχαν αρχίσει ήδη οι παρουσιάσεις ε, προς το συνάδελφο από την Τσεχική Δημοκρατία θα θέσω τα ερωτήματά μου, αλλά ίσως μπορεί να απαντηθούν και από κάποιους άλλους προσκεκλημένους, αν θέλουν. Όσον αφορά το θέμα που θέσατε για την εκ των προτέρων ερεσιμότητα στο πλαίσιο της γραφειοκρατίας και ότι χρειαζόμαστε απλοποίηση, πολύ σωστό είναι αυτό, αλλά στην παρουσίασή σας είπατε επίσης το εξής, ότι ένας μεγάλος αριθμός οργανισμών και φορέων συμμετείχαν ε, και αυτό είναι σφάλμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ή εσείς ως κράτος μέλος θα μπορούσατε να απλοποιήσετε ε, την κατάσταση. Δεν είναι μόνο λάθος Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είναι και πολλά που μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν για να είναι απλούστερο το σύστημα. Θα ήθελα απλώς να κάνω ένα σχόλιο ως προς αυτό. Δεύτερον, η παρακολούθηση των ερεσιμοτήτων των εκ των προτέρων. Εξηγήσατε την κατάσταση και το σύστημα στην ε, Τσεχική Δημοκρατία όμως. Μερικές φορέ, η εσωτερική παρακολούθηση είναι πράγματι αποτελεσματική. Μερικές φορέ, γιατί το, η κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του κράτους μέλους δεν θέλουν να επικρίνουν την απόδοσή τους ε, ε, ε, γι' αυτό ίσως ε, θα ήταν καλύτερο να είναι εξωτερική η παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας των ερσιμοτήτων αυτών. τρίτων. όσον αφορά στις κυρώσεις, αναφέρατε στην παρουσίασή σας ε, ότι δεν πιστεύετε ότι ε, ε, δεν θα έπρεπε να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει αναστολή πληρωμών ή κυρώσισμα δεν υπάρχει, αν, δεν, αν δεν γίνεται αυτό, δεν υπάρχει λόγος να έχουμε και εκ των προτέρων ερεσιμότητες. Εσείς, αν δεν συμφωνείτε με αυτές τις αναστολές ή τις κυρώσεις, τι ακριβώς θα προτείνατε σε περίπτωση μη πλήρωσης των ερεσιμοτήτων. Πρόεδρο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ζητήσω τώρα από του προσκεκλημένους να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Έχετε 10 με 15 λεπτά στη διάθεσή σας, ε, όλοι μαζί. Ποιο θέλει να ξεκινήσει. Κύριε Καθηγητά, Μία από τις ερωτήσεις που κάνατε στην αρχή μας είπατε αν μπορούμε να πούμε ότι εκ των προτέρων ε, ρεσιμότητες είναι ε, εγγύηση για την επιτυχία. Όχι είναι η απάντηση, όμως είναι πάρα πολύ σημαντικό για να τεθούν τα θεμέλια. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ως προς αυτό. Τις χρειαζόμαστε. Το επόμενο ερώτημα ήταν πώς μπορούμε να τις καταστήσουμε πιο αποτελεσματικές οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα πρόβλημα λιγότερο από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν πρέπει να υπάρχει υποψία διάκριση κατά ε, κάποιου κράτου μέλους. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν λιγότερο ε, αυτό το πρόβλημα, δεν έχουν αυτό το πρόβλημα και έτσι υπάρχουν κάποιε ημερομηνίε εκπνοή. Αν μία μέχρι συγκεκριμένη ημερομηνία δεν πληρωθούν οι ε, προποθέσει. τότε πρέπει να δώσει κανείς πίσω τα κονδύλια. Και αυτό επισπεύδει τη διαδικασία γιατί κάποιοι άλλοι περιμένουν ήδη για να ε, ε, προσχωρήσουν. Επίσης, ε, λειτουργούν με ε, διαπιστευμένες οργανώσεις. Εντάξει, δεν μπορεί να το κάνει αυτό κανείς με τις κυβερνήσεις, αλλά ε, στην περιφερειακή πολιτική μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος. Είναι προϋπόθεση το να δουλεύει κανείς με εξουσιοδοτημένους, διαπιστευμένους φορείς. Είναι όχι εγγύηση, αλλά είναι μια ευνοϊκή προϋπόθεση για να επιτύχει η εφαρμογή ενός προγράμματος. Αυτό κάνουν οι Αμερικανοί και ειδικότερα όσον αφορά την ημερομηνία εκπονοής, το sunset date όπως το αποκαλούν, ε, εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ελκυστικό. Ευχαριστώ. Ποιος θα συνεχίσει? Κυρία Ντουπρέ. Ο Τσέχος συνάδελφος τότε. Α, ναι, θα προσπαθήσω να απαντήσω στην τελευταία τελευταία ερώτηση που θέσατε. Όσον αφορά την απλούστευση και τον αριθμό των ε, συμμετεχόντων ε, φορέων, η απάντηση είναι ναι. Η τσεχική δημοκρατία, η... τα θεσμικά χαρακτηριστικά της ε, είναι αρκετά περίπλοκα. Έχουμε πολλά υπουργεία και πολλούς κρατικούς ε, φορείς. Η κατάσταση είναι πολύ πιο περίπλοκη και δυσκολότερη όταν πρέπει να εξευρεθεί μια λύση σε εθνικό επίπεδο. Αλλά και κατά δεύτερον, ε, η δημιουργία ολόκληρης της έννοιας των εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων είναι πάρα πολύ περίπλοκη, οπότε δημιουργεί ένα περιβάλλον ε, που δεν ευνοεί την εύκολη εξέβρεση λύσεων, αν με καταλαβαίνετε. Ε, η τέλεια λύση, εμπροκειμένο, θα ήταν να μην έχουμε εκ των προτέρων αιρεσιμότητες ή να γίνονται διαπραγματεύσεις ε, με τα κράτη-μέλη να βλέπει κανείς τα ισχυρά και τα αδύναμα του σημεία ε, και να ε, τίθενται επιτάπητος ε, συγκεκριμένες εκ των προτέρων αιρεσιμότητες για το συγκεκριμένο κράτος μέλος. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια, αλλά για το μέλλον κατά τη γνώμη μας είναι η καλύτερη λύση. Αν υπάρχουν αν, υπάρχει μία, ένα πρόβλημα, ε, καλό θα ήταν να γίνουν διαπραγματεύσεις ε, ε, καλύτερες και επαρκέστερες με τα κράτη-μέλη, ώστε να υπάρχουν εκ των προτέρων ερεσιμότητες που θα είναι πιο στοχευμένες και που θα αμβλύνουν σε ανησυχίε των κρατών μελών. Αυτή είναι η απάντησή μου λοιπόν σε σχέση με την απλούστευση, την απλοποίηση. Όσον αφορά τώρα τις κυρώσεις που, μας, που αναφέρατε. Κοιτάξτε, αν υπήρχε μικρότερος αριθμός εκ των προτέρων ερεσιμοτήτων και συζήτηση στο πλαίσιο της πρότασης του κανονισμού, ε, και υπήρχε αποδέσμευση των κονδυλίων εγκαίρων, θα μπορούσαμε να βρούμε τρόπους αντιμετώπισης ακόμη και πριν από το στάδιο της εφαρμογής. Γιατί τώρα βρισκόμαστε σε μια κατάσταση ε, εφαρμογής προγραμμάτων και έργων χωρίς να πληρούνται όλες οι αιρεσιμότητες και αυτό είναι επικίνδυνο για τα κράτη-μέλη γιατί επενδύουμε εκ των προτέρων πολλά, αλλά απ' την άλλη δεν είμαστε πάρα πολύ βέβαιοι κατά πόσο θα υπάρχει αναστολή πληρωμών ή όχι. Ε, όσον αφορά λοιπόν ε, το φιλοσοφικό επίπεδο, εν πάση περιπτώσει, ίσως ε, να μην τίθενται οι κυρώσεις ως βασικό σημείο κατά τη διάρκεια της συζήτησης. Η κυρία Ντεπρέ. Είναι παρεμβάσει οι οποίε έθιξαν το ζήτημα τη περιπλοκότητας και την ανάγκη της απλούστευσης στο ζήτημα της αιρεσιμότητα. Εάν δούμε τις διεθνείς εμπειρίες του Διεθνού Νομισματικού Ταμείου και άλλων, αυτή η ήταν και η τάση τα τελευταία χρόνια, προσπαθήσουν να περιορίσουν τον αριθμό των αιρεσιμοτήτων. Δεν είναι τόσο απλό στην πράξη, διότι οι προθέσεις ε, ε, είναι καλές. Δεν λένε, λένε συνεχώς ότι θα περιορίσουν τι αιρεσιμότητες, αλλά στην πράξη βλέπουμε ότι υπάρχει ένα χάσμα. Παρά τα αυτά όμως ε, υπήρξε ένα κίνημα και μια κίνηση προς ε, μια μείωση τα τελευταία αυτά πέντε χρόνια. Αυτό που έχει σημασία είναι να μην ε, επανεφεύρουμε τους κανόνες κάθε φορά, διότι μιλάμε για οικοδόμηση ικανοτήτων για την εφαρμογή αυτών των ερεσιμοτήτων. Χρειάζεται πολλή χρόνο. Εάν λοιπόν οι κανόνες τροποποιούνται συχνά, επανεφεύρονται σε κάθε προγραμματική περίοδο, αυτό προκαλεί πολλές επιπλοκές ε, για τις τοπικές αρχές, ε, για τα κράτη, προκειμένου να μπορέσουν να τις εφαρμόσουν. Τώρα σε επίπεδο ανακοίνωσης πώς θα διαδώσουμε τις βέλτιστες πρακτικές είναι κάτι το οποίο γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στην Ευρώπη. Δεν έχουμε πολλές ανακοινώσεις ε, πάνω στο θέμα, δηλαδή πλατφόρμες όπου στην ουσία μπορούμε να μάθουμε τις νέες ε, και βέλτιστες πρακτικές, πώς οι δικαιούχοι μπόρεσαν να προχωρήσουν, να υποφεληθούν από αυτές τις βέλτιστες πρακτικές. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει και που υπάρχει και σε άλλα κράτη του ΩΣΑ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριο Μπέρκοβιτς, την Κομισιόν. Ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, αλλά ελπίζω σαφής. Μου άρεσε πολύ η περιγραφή του κυρίου Ολμπρεχτ. Η μία πτυχή είναι η αποτελεσματικότητα η εφαρμογή οι προϋποθέσεις ε, ε, εκ των προτέρων ε, μας δείχνουν ότι θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν αποτελεσματικά και αυτός είναι ο καλύτερος τρόπος για να δούμε το ζήτημα τώρα στο, το θέμα των προθεσμιών του διοικητικού άκου και ούτω καθεξής. Είναι πολύ επικίνδυνο να συζητήσουμε αυτά τα θέματα μεμονωμένα. Υπάρχουν ε, καθυστερήσεις στην ε, απαρχή προβλημάτων, την εκταμείευση κλπ. Αλλά σύμφωνα με τις εκ των αυτό είναι ένα μικρό στοιχείο, μικρός παράγοντας σε ό,τι φορά το ζήτημα του, της ανάθεσης. Πολλά αυτά τα στοιχεία προς το παρόν δείχνουν ότι είναι πολύ σημαντικά, αλλά υπάρχουν σημαντικότερα ζητήματα Γι' αυτό λοιπόν αυτού του είδους συζητήσεις θα πρέπει να βάλουν νομού όλα τα στοιχεία και να συναντάγουν ποιε είναι οι πραγματικές αιτίε. Με τα χαρά να τους συζητήσουμε περαιτέρω το θέμα. Τώρα σε ό,τι αφορά τον βαθμό της ε, εκπλήρωσης ε, αυτό που σας παρουσίασα ήταν μια εικόνα στα μέσα του 2015. Τα πράγματα προόδευσαν, σημαντικά. Και εκεί θα εστιάσει και η έκθεση την οποία ανέφερα στην παρέμβασή μου. Το ζήτημα της τεχνικής ε, βοήθειας υπάρχει μια ιστορία για το θέμα της ε, των προτέρων αιρεσιμότητας. Χρειάζεται ικανότητα σε όλα τα επίπεδα και η τεχνική βοήθεια είναι διαθέσιμη σε όλα τα επίπεδα έχουμε καταδείξει από πλευρά της Κομισιόν ότι η τεχνική βοήθεια μπορεί να χορηγηθεί προκειμένου να ε, εκπληρωθούν οι εκ των προτέρων αιρεσιμότητες. Τώρα σε ό,τι φορά το ερώτημα του κ. Βανλίστερου, συμφωνούμε απόλυτα μαζί σα. Τώρα είναι η ώρα να δείξουμε τα θετικά χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής. Θα εκδώσουμε διάφορα έγγραφα να σας πω ότι θα υπάρξει ένα έγγραφο για τις εκ των προτέρων θα υπάρξει επίσης και μια ανακοίνωση για την ε, ευφυή εξειδίκευση. Ε, υπάρχουν λοιπόν διάφορα στοιχεία τα οποία θα μπορέσουν να εξηγήσουν τα θετικά χαρακτηριστικά αυτής της πολιτικής σε ό,τι φορά το θέμα κατά πόσον αυτό υπονομεύει τις ε, περιφερειακές ιδιαιτερότητες δεν υπάρχει τέτοια απόδειξη για την υποβάθμιση των, διο... Ε, των περιφερειακών ιδιαιτεροτήτων ε, του αντίον ε, το θέμα της ευθύους εξειδίκευσης είναι κάτι το οποίο οθεί σε περαιτέρω εξειδίκευση. Θα υπάρξει μια προσέγγιση από την ε, βάση στην κορυφή και όχι το αντίστροφο θέσατε και μια ερώτηση που αναφερόταν στις ε, τσεχικές αρχές. Ε, κάτι το οποίο ήταν χρήσιμο για αυτές τις ε, ρεσιμότητες κατέληξε την περιπλοκότητα που υπάρχει σε κάποια κρατημέλη και η δυσκολία σε ό,τι αφορά το συντονισμό μεταξύ των διαφόρων οργάνων. Και αυτό οδήγησε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν πώς θα οργανώσουν την διαδικασία, να ενισχύσουν τον ρόλο των κεντρικών συντονιστικών οργάνων το ότι, ε, μόνο το ότι υπάρχουν τόσε ε, πολλά όργανα που εμπλέκονται, αυτό οδήγησε σε ε, δημιουργία δυσκολιών. Αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία. Τέλος, σε αυτή τη γενική ερώτηση για την ε, δεξορθολογισμό της εκ των προτέρων αιρεσιμότητας, νομίζω ότι στόχο τη της αιρεσιμότητας ήταν να φτάσουν σε ένα κάποιο επίπεδο τώρα και το πολύ μέχρι τα τέλη του έτους όλοι θα πρέπει να πληρούν αυτές τις αιρεσιμότητες. Το θέμα είναι τι περιεχόμενο παρέχεται σε αυτές και δίνεται σε αυτές τις ε, εκ των διότι δεν θα διατηρηθούν οι ίδιες εάν πρόκειται να μην εκπροθούν αλλά ταυτόχρονα δεν θα εφεύρουμε και νέε αρεσιμότητε που θα πάνε κάτι πέρα από, από το λογικό από το εύλογο Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για το ενδιαφέρουσα, ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις και για τη συζήτηση. Ολοκληρώθηκε το σημείο αυτό της ημερησίας διατάξεως. Ευχαριστώ κυρία μου, κύριοι μου. Ίσως να έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε εδώ στην Επιτροπή Ρέτζο και προχωράμε στην ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο κυρία Κρέτσου η οποία θα έπρεπε να έχει φτάσει. Δεν ξέρω. I Ladies and gentlemen, can I ask you to take your seats? Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Και σας παρακαλώ ησυχία στην αίθουσα. Can we continue now? Thank you very much. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούμε τώρα να συνεχίσουμε με την ανταλλαγή απόψεων με την Επίτροπο Κορίνα Κρέτσου, Επίτροπο Περιφερειακής Πολιτικής και Πολιτικής Συνοχής για τα κυριότερα σημεία του 2016. Η Επίτροπος κυρία Κρέτσου έχει έρθει στην Επιτροπή μας για μια ανταλλαγή απόψεων τρεις φορές φέτος ήδη τον Ιανουάριο, τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. Και σήμερα έχει έρθει στην Επιτροπή μας για να κάνουμε μία ανασκόπηση του 2016 των σημαντικότερων γεγονότων και να δούμε τι μας περιμένει το 2017, τι περιμένει την Ευρωπαϊκή Περιφερειακή Πολιτική το επόμενο έτος. για την Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης κυριότερες στιγμές του 2016 ήταν τα τόπα για την Ελλάδα και την Κύπρο και η πρώτη ενταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 23, την περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας αν θυμάστε. Επίσης, εγκρίθηκαν 8 μη νομοθετικές εκθέσεις το 2016, ολοκληρωμένες ε, εδαφικές επενδύσεις, εργαλεία περιφερειακής ανάπτυξης, πολιτική συνοχή, ε, κυρία Γιώτοβα, Τόμασιτς, ε, την εξειδίκευση, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της κυρίας Ντομάτο, έκθεση για την στρατηγική των Άλπαιων της κυρίας Μπρέσο, Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία της Υποφαινόμενης και Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλληλεγγύης του κυρίου Τσίκο. Σήμερα θα ψηφίσουμε για την έκθεση σχετικά με το άρθρο 16, εφαρμογή της πολιτικής συνοχής το 2014 και 2015, την έκθεση του κυρίου Βανίστελ Ρόι. Πρώτο μέλημά μας του χρόνου θα είναι η συνέχεια της συζήτησης για το πρόγραμμα διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων υπό την Μαλτέζικη Προεδρία και θα συζητήσουμε την πρόταση Omnibus. Και θα συνεχίσουμε την συζήτηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το πρόγραμμα εργασίας του 2017. Επίσης υπάρχει και η ανακοίνωση για την ευφυή εξειδίκευση και την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την επόμενη φάση της πολιτικής συνοχής. Έχουμε λοιπόν πολλά να πούμε σήμερα με την Επίτροπο και θα ακολουθήσω την ε, συνήθισμένη διαδικασία. Θα ακούσουμε την ε, Επίτροπο κυρία Κρέτσου, μετά θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε ερωτήσεις, πρώτοι συντονιστές των πολιτικών ομάδων και έπειτα οι υπόλοιποι. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στην Επιτροπή σας. Ε, κυρία Πρόεδρε, κύριε Μιχαήλουβα, αγαπητοί συνάδελφοι, καλημέρα σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Όπως γνωρίζετε χαίρομαι πάντα κάθε φορά που έρχομαι στην Επιτροπή σας, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης και παρά το γεγονός ότι ήδη έχουμε συναντηθεί αρκετές φορές μέσα στο 2016 θα ήθελα να λάβω την ευκαιρία για να κάνω μια ανασκόπηση των κυριότερων στιγμών του έτους. Όπως είπε η κυρία Πρόεδρος, περνάμε δύσκολες ε, εποχές και έχουμε όντως πάρα πολλά να πούμε. Ίσως θα γνωρίζετε πως έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα από την τελευταία φορά που συναντηθήκαμε. Έχουμε πολλές εξελίξεις παγκόσμια και πιστεύω πως ε, αυτή η συζήτηση θα είναι λίγο πιο πολιτική. Θα συζητήσουμε για το τι θα θέλαμε να έχουμε από την ε, πολιτική μας ε, η περιφερειακή πολιτική έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια και αλλάζει συνεχώς. Και όπως ξέρετε η περιφερειακή πολιτική και η πολιτική συνοχής ε, δεν ήταν πάντα κάτι το εύκολο. από την δημιουργία το 1968 της Γενικής Διεύθυνσης για Περιφερειακή Πολιτική μέχρι την ε, αλλαγή του 1974 και τον κανονισμό που εγκρίθηκε το 1975 για την πολιτική συνοχής ε, βρισκόμασταν συνέχεια υποδρυμία κριτική. Τώρα όμως είναι πολύ σημαντικό, πιο σημαντικό από ποτέ να συζητήσουμε την ε, ε, περιφερειακή και πολιτική και την πολιτική συνοχή Και ε, ξέρετε ποιο ήταν ο πρωτεργάτης, ο George Thompson, Βρετανός, όσο ειρωνικό και αν ακούγεται αυτό. Και μάλιστα στην έκθεσή του είχε γράψει, ο, ε, ήταν μια έκθεση ε, πάρα πολύ γνωστή, είχε γράψει λοιπόν ο κύριος Τόμσον ότι καμία κοινότητα δεν μπορεί να διατηρήσει την ύπαρξή της, δεν μπορεί να συντηρήσει τους πολίτες εάν δεν υπάρχει συνεργασία. Υπάρχουν πολλές διαφορές ανάμεσα στις περιφέρειες, πολλά, ε, πολλές διαφορές στο βιωτικό επίπεδο και η συνεργασία λοιπόν και η συνοχή είναι η καλύτερη λύση. Ε, πάλεψε λοιπόν για την δημιουργία της ε, πολιτικής περιφερειακής ανάπτυξης. Όπως ξέρετε, το 1974 υπήρχαν μεγάλες εντάσεις. Η Ιταλία και η Μεγάλη Βρετανία απείλησαν να μην συμμετέχουν σε μελλοντικές συνεδριάσεις του Συμβουλίου εάν δεν προχωρούσε η πολιτική περιφερειακής ανάπτυξης. Ε, γι' αυτό λοιπόν και τότε δημιουργήθηκαν τα θεμέλια της ε, πολιτικής με στόχο να μειωθούν οι ε, ανισότητες ανάμεσα στις διάφορες περιφέρειες, τις περισσότερο και τις λιγότερο ανεπτυγμένες. Και όπως είχε πει ο κύριος Τόμσον τότε, ήταν μια ηθική, ε, ήταν ένα ηθικό καθήκον να γίνει αυτό. Η πολιτική μας λοιπόν έχει περάσει από πολλά στάδια, έχει υποστεί πολλές αλλαγές από τότε μέχρι τώρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτή τη στιγμή βρίσκεται ενώπιον τεράστιων προκλήσεων. Είναι μία προειδοποίηση, ένα καμπανάκι αν θέλετε. Οι περιφέρειες της Ευρώπης έχουν και αυτές αλλάξει, αλλά έχει αλλάξει και ο τρόπος ανάλυσης μας. Είμαστε απόλυτα ενήμεροι για τις ε, προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει μια πολύ εύθραυστη οικονομική ανάπτυξη. Είναι Ηράκλειο το έργο της ε, προσπάθειας για επανένταξη στην αγορά εργασία εκατομμύριων νέων ανέργων. Υπάρχουν εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες που ζουν στα όρια της φτώχειας και υπάρχει τεράστια ανάγκη για αλληλεγγύη αλληλεγγύη ε, προ τα άτομα που απειλούνται από την πείνα, την ανεργία, την ε, ένδυα. Υπάρχουν επίσης και μεγάλες διαφορές ανάμεσα στα κράτη-μέλη και αυτές οι διαφορές διαβρώνουν τα θεμέλια του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Επίσης ε, νιώθουμε την ανασφάλεια. Είναι αισθητή. Αυτή η ανασφάλεια μας οδηγεί σε φόβο και σε υπονόμευση τη Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη πάνω στην οποία στηρίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δίχως αμφιβολία πρέπει να είναι κοινό μας στόχο να βελτιωθούν αυτές ε, οι συγκυρίες. Και είμαι απόλυτα πεπισμένη ότι ακριβώς σε τέτοιες, σε τόσο δύσκολες στιγμές η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλήσεις των πολιτών, στις προκλήσεις ανεξάρτητα από το πού διαμένει ο κάθε πολίτης. Όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να είναι σε θέση να υποφελούνται από την ε, Ένωση και να έχουν ίση πρόσβαση στις ευκαιρίες. Αυτό σημαίνει πολιτική συνοχής. Είναι εξίσου όμως σημαντικό η πολιτική συνοχής να είναι χωρίς αποκλεισμού, να ε, εισακούει τις ανησυχίες των πολιτών, να δημιουργεί ε, συνέργειες, συνεργασίες ανάμεσα σε άτομα, κυβερνήσεις, περιφέρειες είναι πολύ σημαντικό, όσο, δύσκολος, όσο δύσκολο και αν είναι, να υπάρχει ένας διάλογος, έτσι ώστε να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη, να ενισχυθεί η συνεργασία και η συνεργασία μάλιστα για έναν κοινό στόχο. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη φάση, στο στάδιο συζήτησης του επόμενου προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι κάτι τεχνικό. Η συζήτηση που θα προηγηθεί θα είναι πολιτική. Θα ε, συζητηθούν οι θεμελιώδεις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει να δούμε πώς θα βελτιώσουμε την πολιτική συνοχή, πώς θα ε, την προσαρμόσουμε και σίγουρα θέλει βελτίωση, βελτίωση και στις λεπτομέρειες. Πρέπει λοιπόν να είμαστε σε ετοιμότητα έτσι ώστε να μην διακινδυνεύσει η κατάρρευση του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Από την αρχή της θητείας μου ε, συνεργαζόμουν και συνεχίζω να εργάζομαι για τους ε, στόχους αυτούς. Έχουμε εργαστεί πάρα πολύ σκληρά με τα κρατημέλη και με τις περιφέρειες για να ολοκληρώσουμε με επιτυχία το προηγούμενο πρόγραμμα και να επιταχύνουμε την ε, δρομολόγηση του επόμενου έχουμε ε, δώσει έμφαση στις πιο φτωχές περιφέρειες. Δεν θέλω βέβαια εδώ να κατονομάσω ή να ασκήσω κριτική, αλλά χρειάζεται να βρούμε πολύ συγκεκριμένες λύσεις για πολύ συγκεκριμένα προβλήματα. Έχουμε εργαστεί επίσης πάρα πολύ σκληρά για να συμπεριληφθούν και οι πόλεις στην ε, υλοποίηση της ε, περιφερειακής πολιτικής. Και με χαρά μου παρουσίασα τον οκτώ. Οκτώβρη στο στα πλαίσια των ε, ε, Ηνωμένων Εθνών το νέο αστικό θεματολόγιο που ε, δημιουργήθηκε, που μάλλον τέθηκε σε ισχύ από την Ολλανδική Προεδρία. Στόχος μας είναι να διορθώσουμε τις αδυναμίες μας και να ενισχύσουμε τα καλά μας στοιχεία. Πρέπει επιτέλους να δείξουμε τι σημαίνει πολιτική συνοχή, σημαίνει δημιουργία θέσεων απασχόλησης, σημαίνει δημιουργία κατάλληλων υποδομών στις πόλεις για να ευνοηθεί ανάπτυξη και στις περιφέρειες επίσης. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι δεν είναι όλα ρόδινα. Φυσικά και υπάρχουν προβλήματα, φυσικά και πρέπει να συνεχίσουμε τι πιέσει στι κυβερνήσει και στι περιφερειε για να επιταχύνουν την υλοποίηση των προγραμμάτων περιφερειακή πολιτικής. Χρειάζεται καλύτερη συνεργασία με του υπουργού και χρειάζεται η συμμετοχή δική σας τόμε και από εσάς για να μπορέσετε να μεταδώσετε αυτό το μήνυμα στις περιφέρειές σας. Έχουμε επικαιροποιήσει τους ε, σχετικούς κανονισμούς και σε συνεργασία με τον Επίτροπο Κάλλα και προσπαθούμε να ακούσουμε με μεγάλη προσοχή τις ανησυχίες των πολιτών για αυτές τις πολιτικές. Γι' αυτό λοιπόν ε, ε, ελπίζω στην στήριξή σας την, το επόμενο έτος, το 2017, όταν θα έρθει η ώρα έγκρισης της νέας πολιτική. Φυσικά και μπορούμε να ασκήσουμε ε, πολύ μεγάλη κριτική στα προβλήματα που υπάρχουν. Χρειάζεται σίγουρα πλούστευση, χρειάζεται μεγαλύτερη σχέση με τα προβλήματα των ε, πολιτών. Αλλά, αγαπητοί ευρωβουλευτές, πρέπει να έρθει η ώρα να εφαρμόσουμε τα ευρωπαϊκά προγράμματα, να εφαρμόσουμε προγράμματα τα οποία θα δίνουν έμφαση στις ε, τοπικές ε, κοινότητες και θα βοηθήσουν όλους τους πολίτες. Έχει έρθει η ώρα να γίνουμε πολύ πιο δημιουργικοί στο πώς ενημερώνουμε και πληροφορούμε τους πολίτες για την περιφερειακή πολιτική. Αυτό είναι κάτι στο οποίο έχουν παρατηρηθεί μεγάλες ελλείψεις και πρέπει να το διορθώσουμε. Και εδώ Πάλι θα αναφερθώ σε εσά ως πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία ε, για την επιτυχία αυτή ε, ενημέρωση των πολιτών. Διότι, όπως γνωρίζετε, η πολιτική συνοχή ε, είναι μια ευρωπαϊκή υπόθεση, είναι ένα στίχημα που πρέπει να κερδίσουμε και είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να μεταφέρει σε κάθε γωνιά της Ευρώπης τα ευρωπαϊκά ιδεώδη και να δώσει στα παιδιά μας ένα καλύτερο μέλλον. Όπως σας είπα, ε, αφιερώνω από την αρχή της θητείας μου και θα αφιερώνω όλη μου τη δύναμη για να προωθήσω τις ε, καλές συνέργειες, αλλά όπως σας είπα και πριν, είναι κοινή η προσπάθεια. Ελπίζω λοιπόν στη δική σας στήριξη, στη δική σας βοήθεια για να μεταδώσετε τα ε, αποτελέσματα και τις επιτυχίες της περιφερειακής πολιτικής σε κάθε γωνιά της Ευρώπης. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ξεκινήσουμε με τον πρώτο γύρο ερωτήσεων και σχολείων από τους συντονιστές. Ο κύριος Όλμπιτ ε, από το ΕΛΚ. Κυρία Επίτροπε, νομίζω ότι τρία στοιχεία θα ήθελα να αναφέρω και να σας ρωτήσω. Υπάρχει το χθες, το σήμερα και το αύριο. Εχθές ε, είχαμε ε, ε, επειδή αναφερθήκατε στο Ηνωμένο Βασίλειο, είχαμε τη συζήτηση για το τι θα έπρεπε να είναι η πολιτική συνοχής. Ε, μείωση των ανισοτήτων, μετά είχαμε τη λισαβονοποίηση η λισαβονοποίηση ήταν μια πολιτική συνοχή πολύ περισσότερο υπέρ της ανάπτυξης και σήμερα συνεχίζουμε και τα δύο. Και μείωση των ανισοτήτων και την ανάπτυξη σε, όλες τις, όλα τα κράτη-μέλη. Ε, θέλουμε ανάπτυξη, αλλά όχι μόνο για τους πιο αδύναμους. Τώρα έχουμε ένα πολύ χαμηλό ποσοστό εφαρμογής. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όταν συζητούμε λοιπόν την κατάσταση, νομίζω, επειδή το συζητήσαμε πριν από 10 λεπτά για ένα άλλο θέμα, πρέπει να τονίσουμε την πραγματική προέλευση ε, των αιτίων της, της, ε, του χαμηλού επίπεδου εφαρμογής. Είναι πρόβλημα νομοθεσίας, είναι πρόβλημα των κρατών μελών, είναι πρόβλημα ε, των ευρωπαϊκών θεσμών, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί... Έχουμε φτάσει ήδη στο τρίτο έτος και το επίπεδο εφαρμογής σε μερικές χώρες ε, είναι 0%. 1% στη δική μου χώρα. Ε, είναι ε, γεγονός ότι αυτό δημιουργεί μια διαφορετική προσέγγιση για τους καθαρούς εισφορείς και ξέρετε πολύ καλά ότι, πρέπει, ότι θέλουν να ε, μειώσουν, να πάνε προς τα πίσω και να ε, ζητούν μόνο τη μείωση των ανισοτήτων και να μην υπάρχει καμία αναφορά στην ανάπτυξη. Ε, πολύ ε, λιγότερα χρήματα λοιπόν στην πολιτική συνοχή, πώς μπορούμε να αλλάξουμε δηλαδή τον προϋπολογισμό ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης με όλα τα εξωτερικά στοιχεία που είναι εκτός του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού, για να μπορέσουμε να έχουμε δηλαδή πραγματικά αποτελέσματα με την πολιτική ε, ε, συνοχή και το πρόβλημα των καθυστερήσεων μέχρι το 2020. Χρειαζόμαστε περισσότερα χρήματα για την πολιτική συνοχή για τα επόμενα χρήματα και για τα επόμενα χρόνια και λιγότερα χρήματα για άλλα θέματα όπως για παράδειγμα η μετανάστευση και το ξέρουμε. Ναι, θα είναι χαμηλά την επόμενη χρονιά, αλλά τη μεθεπόμενη χρονιά θα ε, αυξηθεί. 18, 19, 20 λοιπόν έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση. Μπορούμε να υπερασπιστούμε τις επιλογές μας για την περίοδο αυτή και πολλοί συνάδελφοι είναι εντελώς κατά της πολιτικής συνοχής ε, και αυτό είναι μία τάση κατανομή των ίδιων κονδυλίων σε διαφορετικές ε, γενικές διευθύνσεις Ευρωπαϊκής Επιτροπής να περάσουν κάποια από διαφορετικές γενικέ διευθύνσεις. Το ξέρετε πολύ καλά αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο. Χρειάζεται περισσότερη επικοινωνία για το τι είναι η πολιτική συνοχή. Ξέρουμε τι είναι η πολιτική συνοχή για το μέλλον. κάνουμε αυτή τη συζήτηση, πρέπει να την κάνουμε στην Επιτροπή μας, ε, γιατί έρχεται αυτή η συζήτηση, πλησιάζει με βήματα γοργά και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε. Υπάρχει μια πραγματική ανάγκη επίγουσα να συζητήσουμε το μέλλον της πολιτικής συνοχής και να απαντήσουμε, να απαντήσουμε το ερώτημα θέλουμε ανάπτυξη ή θέλουμε επιστροφή πίσω απλώς στην ε, απλή ε, ε, μείωση των ανισοτήτων. Θέλει να το έχουμε αυτό ενσωματωμένο στην Γενική Διεύθυνση Περιφερική ανάπτυξης μόνο ή θέλουμε να είναι ε, σε όλες τις γενικές διευθύνσεις ε, κατακαιρματισμένο ε, και να προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να το περάσουμε. Είναι δύσκολη αυτή η στιγμή, είναι δύσκολη η στιγμή γιατί δεν είναι μόνο ζήτημα στιγμή προώθησης της πολιτικής συνοχής αλλά αναδιάρθρωσης και πολύ προσεκτικού σχεδιασμού για το μέλλον γιατί είναι μια δύσκολη χρονική συγκυρία αυτή και του χρόνου ενδεχομένως να είναι η πιο σημαντική χρονιά για τη συζήτηση της πολιτικής συνοχής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Φέστβα, λεκμερούς των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, θα ήθελα να αναφερθώ στην πολιτική συνοχή και ε, το κάνω τώρα γιατί πρέπει να παρουσιάσω μια έκθεση μια άλλη επιτροπή αργότερα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε εδώ. Έχετε μια πολύ καλή σχέση με την επιτροπή μας ε, και αυτό φαίνεται γιατί έχετε πάρα πολύ παλιές και καλές σχέσεις με το Κοινοβούλιο. Καταλαβαίνετε το έργο μας, ήσασταν κι εσείς άλλωστε εδώ και όλοι αναγνωρίζουμε την ε, σκληρή δουλειά που έχετε κάνει. Θα ήθελα ε, να πω πως αρχίσαμε να μιλάμε τελευταία για αλληλεγγύη και γιατί από τη μία, τα ταμεία, από την άλλη η πολιτική συνοχή ε, υπήρχε ανάγκη να δημιουργηθούν. Όπως είπε και ο κύριος Όλμπριχτ, η αλληλεγγύη δεν είναι μονόδρομος. Η αλληλεγγύη σημαίνει ε, μαζί, όλοι μαζί, συνεργασία. Ο κύριος Όλμπριχτ ήταν ε, συντάκτης της ε, σχετικής έκθεσης και πιστεύω πως είχε κάνει εξαιρετική δουλειά ε, για το για το να έχουν όλες οι περιφέρειες της Ευρώπης ίση πρόσβαση στην χρηματοδότηση. Ιδιαίτερα για συγκεκριμένες περιφέρειες, μεταβατικές περιφέρειες όπως λέγονται. Καταφέραμε λοιπόν να, εφαρ... να εφαρμόσουμε τις θέσεις μας και να πω ότι υπάρχουν πολλέ διαφορέ. Στη Γερμανία, για παράδειγμα, υπάρχει μια περιφέρεια, η Βαβαρία, η οποία είναι από τι πιο πλούσιε περιφέρειες τη Ευρώπη. Ωστόσο, μέσα σε αυτή την ε, περιφέρεια υπάρχουν ορισμένε, περιοχές οι οποίε ανήκουν στι φτωχότερε τη Ευρώπη. Αυτό πιστεύω ήθελε να πει και ο κύριος Όλμπριχτ όταν μιλούσε για ανισότητες και για διαφορέ. Και αυτό βέβαια δεν είναι ένα πρόβλημα που, πρέπει και που μπορεί να το λύσει μόνο το Κοινοβούλιο ή μόνο η Κομισιόν. Χρειάζονται πολιτικοί οι οποίοι θα εκπροσωπούν τις περιφέρειες, θα εκπροσωπούν τις περιοχές αυτές και ε, θα πρέπει εκείνοι οι πολιτικοί να έχουν απόλυτη επίγνωση του, ε, των αναγκών και ε, που έχει η περιφέρειά τους. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι άνεργοι, χρειάζονται απασχόληση. Από την άλλη όμως πιστεύω πως πρέπει να κοιτάξουμε και τους θεματικούς στόχους και στους θεματικούς στόχους δεν ανήκει μόνο η απασχόληση αλλά και το περιβάλλον για παράδειγμα. Πριν από λίγες εβδομάδες στο Κοινοβούλιο ε, ψηφίσαμε ε, για, ε, τις, για τα περιβαλλοντικά στο ΚΙΤΟ είδαμε κιόλας ε, τη δουλειά που έγινε, συζητήθηκε η κλιματική αλλαγή, το είπατε κι εσείς κυρία Επίτροπα. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ πως είναι απόλυτα αναγκαίο η μελλοντική πολιτική συνοχής και η διαρθρωτική πολιτική να ε, συνεχίσουν να βελτιώνονται, να αναδιαρθρωθούν, διότι κανείς δεν θέλει να δούμε ότι η πολιτική συνοχή και η διαρθρωτική πολιτική θα θυσιαστούν στο βωμό του ΕΦΣΥ έτσι ώστε να διατεθούν από αυτές ε, κονδύλια ε, για, ε, για την οικονομία, για το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Τα χρήματα αυτά προέρχονται από τους Ευρωπαίους πολίτες και πρέπει να διατίθενται πάλι πίσω στους Ευρωπαίους πολίτες έτσι ώστε να πιάνουν τόπο. Ε, υπάρχουν πολλοί τομείς, υπάρχει τεχνολογική ανάπτυξη, υπάρχει ανακαίνιση κτηρίων ε, έτσι ώστε αυτά να καταστούν οικολογικά. Υπάρχουν 8 διαφορετικοί θεματικοί τομείς. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω πως είναι απόλυτα αναγκαίο να έχουμε μια ξεκάθαρη γραμμή την οποία θα ακολουθούμε. Και ανησυχητικό βρίσκω το Συμβούλιο και τις συζητήσεις που γίνονται εκεί. Φοβάμαι πως η φωνή των πολιτών δεν ακούγεται όσο θα ε, έπρεπε ε, εκεί ψηλά. Φυσικά, να πω από την άλλη ότι ο ρόλος ε, των πόλεων είναι πάρα πολύ σημαντικός. Είναι νευραλγική σημασία, θα έλεγα, και πρέπει να φροντίσουμε οι πόλεις να συνεχίσουν να τραβάνε μπροστά την πολιτική συνοχή, αλλά όχι και όχι να υπάρχουν πίσω γυρίσματα. Υπάρχει μία δουλειά, υπάρχει ένα αποτέλεσμα που έχουμε καταφέρει με κόπο να πετύχουμε και πρέπει να προσέξουμε να μην υπάρχει πίσω γύρισμα, να μην οπίστο χωρίσουμε. Αυτό θα θέσει σε κίνδυνο και το ίδιο το ευρωπαϊκό οικοδόμημα. Το είπε και ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου σε μια προηγούμενη ομιλία του εξάλλου. Να επανέλθω λοιπόν στο θέμα. Σίγουρα χρειάζονται πολλές αλλαγές σε πολλά θέματα. Απλούστευση, όπως είπατε και εσείς. Χρειάζεται όμως όχι μόνο απλούστευση, αλλά και να ακολουθείτε η αρχή της συνεργασίας των εταιρικών σχέσεων. Να προσπαθήσουμε να συμπεριλαμβάνονται όλοι οι ε, αρμόδιοι φορείς στη συζήτηση. Και αυτό, ξέρετε, έχει πολλές αντιστάσεις. Αντιστέκονται τα ίδια τα κρατημέλη. Από την άλλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβουλίο και οι Ευρωβουλευτέ και τα κρατημέλη πρέπει να συνεργαστούν και να προσπαθήσουν να προχωρήσουν αυτό το ε, έργο και αυτό γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος, κίνδυνος ε, λαϊκισμού και εξτρεμισμού. Δεν έχουν καμία θέση αυτή στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο που από του Φιλελεύθερου. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήλθατε κύριε Επίτροπε. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξαναβλέπουμε στην Επιτροπή μα και χαίρομαι πολύ που αναφερθήκατε σε πολιτική συζήτηση. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στο μέλλον της πολιτικής συνοχή. Σίγουρα υπάρχουν κίνδυνοι, δεν θα του επαναλάβω, και πρέπει οπωσδήποτε να βρεθεί η κατάλληλη συνταγή, η κατάλληλη αναλογία στη χρήση των ε, κονδυλίων του ΕΦΣΥ, των διαρθρωτικών ταμείων. Ωστόσο, έχω κάποιες ερωτήσεις. Καταρχάς, να πω ότι υπήρξε διαρθρωμένος διάλογος για την περίπτωση της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. Εσείς πώς θα αξιολογούσατε το άρθρο 23 του κανονισμού περί κοινών διατάξεων, πώς ε, θεωρείτε πώς εφαρμόστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποια είναι τα ε, διδάγματα που αντλήθηκαν για το μέλλον της πολιτικής συνοχής. Μετά, οι επόμενες ερωτήσεις μου έχουν σχέση με, τον, με την πρόταση Omnibus. Όπως ε, ξέρετε και εσείς προτείνατε με τους συναδέλφους σας του Σώματος των Επιτρόπων ένα, μια δέσμη μέτρων που θα αφορά το μεταναστευτικό και τους πρόσφυγες. Εσείς πώς σκοπεύετε να ε, αντιμετωπίσετε την διστακτικότητα ορισμένων κρατών για το θέμα αυτό, πώς, ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για την πρόκληση της μετανάστευσης των προσφύγων και ε, τι θα κάνετε με αυτά τα κράτη τα οποία δεν είναι σε θέση, είναι απρόθυμα να υλοποιήσουν τις αποφάσεις για την ένταξη των ε, προσφύγων, την ένταξη, τη στέγαση ε, αυτών των ανθρώπων. Τι σκοπεύετε να κάνετε γι' αυτό. Μετά, άλλη μια ερώτηση σχετικά με αυτό. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να αποτρέψετε τα κράτη-μέλη να υποφελούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, χωρίς όμως να θέλουν να συμμορφώνονται με τους ε, με τους κανόνες, με την ευρωπαϊκή νομοθεσία σχετικά με τους ε, πρόσφυγες, με την ένταξή τους και με τη στεγασή τους. Εγώ θα ήθελα μια πολιτική απάντηση από εσάς για αυτά τα ερωτήματα. Σας ευχαριστώ. Κύριος Λαμαζέ. Κύρια Επίτροπε, ευχαριστούμε πάρα πολύ που αναφερθήκατε ε, σε πολιτικούς όρους σε αυτή τη συζήτηση που είναι πάρα πολύ επίκαιρη, γιατί αυτή τη στιγμή η ανησυχία ε, στο Κοινοβούλιο και στη δική μας Επιτροπή όσον αφορά το μέλλον της περιφερειακής πολιτικής είναι πάρα πολύ έντονη. Και θα ήθελα επίσης να σας ε, ευχαριστήσω γιατί υπενθυμίσατε την ιστορία αυτής της πολιτικής συνοχής που ήταν η πολιτική που επέτρεψε να αντιμετωπίσουμε και να ε, αντιμετωπίσουμε μάλιστα επιτυχώς ε, τις, ε, τα προβλήματα, της της προκλήσεις της περιφερειακής ανάπτυξης. Μπορούμε λοιπόν σήμερα να πούμε ότι έχουμε κάποιες επιτυχίες. Η περιφερειακή πολιτική είναι το κέντρο ε, της ε, ευρωπαϊκής πολιτικής, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πρώτα απ' όλα ένας χώρος αλληλεγγύης. Και νομίζω ότι δεν υπάρχει ε, πολιτική που να την χάνει περισσότερης επίθεσης από ότι η περιφερειακή πολιτική. Παρόλα αυτά όμως δεν υπάρχει και πολιτική που κάνει τόσα πολλά για να ε, αμβλύνει τον πολύ βίαιο χαρακτήρα άλλων πολιτικών που εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πρέπει να, να θέσουμε το ερώτημα της συνοχής των πολιτικών μας. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Όταν από τη μία πλευρά, σε επίπεδο πολιτικής εμπορικής, κάνουμε διαπραγματεύσεις ε, συμφωνιών ελευθέρων συναλλαγών που θέτουν σε ευάλωση τη θέση την παραγωγή μας, που επιδεινώνουν τα ποσοστά ανεργίας στις περιφέρειές μας. Η πολιτική συνοχής παρεμβαίνει λοιπόν για να αμβλύνει τα καταστροφικά αποτελέσματα αυτών των πολιτικών Παράλληλα όμως, οι στόχοι που θέτουμε, οι στόχοι που θέτουμε για την ε, περιφερειακή πολιτική πάντοτε ε, υπαναχωρούν κάπως. Αν για τον, με, τον, με ορίζοντα το 2030, 2050, 190 εκατομμύρια Ευρωπαίοι θα απειλούνται, ε, δεν θα φταίει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα υπάρχει πολιτική συνοχή για να βοηθήσει την κατάσταση, όμως θα είναι και πολύ πιο δύσκολο πλέον να το κάνει αυτό. Δεν επιμένουμε λοιπόν επαρκώς ε, επί των δύο αυτών σημαντικών ε, σημείων της εφαρμογής μιας συνοχής για τις πολιτικές και η δική μας ε, πολιτική συνοχής χα, ε, αμβλύνει σε μεγάλο βαθμό τα καταστροφικά αποτελέσματα πολλών ευρωπαϊκών πολιτικών. Δεύτερη παρατήρηση που θα ήθελα να κάνω είναι η εξής. Γίνεται μια συζήτηση σήμερα θα πάμε προς την επανεθνικοποίηση ή όχι. Θα θέσουμε ένα αμφιβόλο τις κατηγορίες των περιφερειών, θα δημιουργήσουμε ρήξη με τα θεμέλια της πολιτικής μας, δηλαδή την κάλυψη των καθυστερήσεων. Πρόκειται για ζητήματα εξαιρετικά σημαντικά, πολύ πολιτικά, τα οποία χρήζουν, και ξέρω ότι και εσείς συμφωνείτε με αυτό, από σήμερα κιόλα ενό πολύ ενισχυμένου διαλόγου μεταξύ τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή και των μελών τη Επιτροπή Περιφερειακή Ανάπτυξη, ώστε οι προτάσει τι οποίε θα υποβάλουμε και ε, κατά πάσα πιθανότητα ε, μαζί με το Συμβούλιο να είναι οι πιο ε, παραγωγικές. Το 2016 ήταν μία χρονιά κατά την οποία ε, έλαβε χώρα το Brexit με ε, παράλληλα ε, την αναθεώρηση του CSP. Εδώ λοιπόν έχουμε να κάνουμε με ένα ενδεχόμενο Brexit, του κατά πόσο θα αλλάξει το μέσο ΑΕΠ, το, το ΑΕΠ ανα ε, κάτοικο ε, θα υπάρξει και μία μείωση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ήθελα να μάθω κατά πόσο η Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Ανάπτυξης έχει αρχίσει να επεξεργάζεται το ενδεχόμενο του αντικτύπου αυτού και να σας επιστήσω την προσοχή κυρία Επίτροπε, στην ιδιαίτερη κατάσταση της Ιρλανδίας, η οποία θα έχει να αντιμετωπίσει σημαντικές δυσκολίες σε σχέση με αυτό το Brexit και ε, επίσης ε, η διαδικασία της ειρήνης ε, η οποία μπορεί να ε, τεθεί και αυτή ένα αμφιβόλο. Ελπίζουμε ότι η ομάδα μας θα υποβάλει κάποιες προτάσεις που θα μας δώσουν τη δυνατότητα να ε, συνεχίσουμε και να προχωρήσουμε το διάλογο. Για την Επιτροπή μας ένα σημαντικό σημείο ήταν ο διαρθρωμένος διάλογος ε, για τις κυρώσεις κατά της Ισπανίας και της Πορτογαλίας και είμαι πραγματικά ενθουσιασμένος που η Επιτροπή μας και Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, συνέβαλε σε μία λύση που ε, μέχρι σήμερα είναι ικανοποιητική. Πρέπει όμως να σας πω ότι είμαστε και ανήσυχοι ότι γιατί στις 16 Νοεμβρίου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε μία ανακοίνωση σε σχέση με τα ε, σχέδια προϋπολογισμού που αφορούν το, την Κύπρο, το Βέλγιο, τη Φιλανδία, την Ιταλία, τη Λιθουανία και τη Σλοβενία και θα ήθελα και έχουμε μάλιστα ε, και την, το φόβο ε, ότι υπάρχει περίπτωση να ξαναδούμε αυτό το θέμα της αναστολής των κονδυλίων για αυτές τις έξι χώρες που ανέφερα. Το ε, μήνυμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πρέπει να εισακουστεί. Δεν θέλουμε ενεργοποίηση αυτής της διαδικασίας για λόγους ε, αρχής. Ε, όπως ε, σας είπα, ο κανονισμός που πρόκειται να ψηφίσουμε σε σχέση με την τεχνική αρρωγή. Εσείς είστε πολύ δραστήρια όσον αφορά τις άκρος απομονωμένες περιοχές και γνωρίζετε πολύ καλά το ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό ε, και επειδή ε, οι περιοχές αυτές ε, θα μπορέσουν να επωφεληθούν από αυτό αυτές τις ε, πολιτικές θέλουμε να δούμε πώς θα μπορέσει να υπάρξει ένας ε, μηχανισμός τεχνικής αρρωγής ενισχυμένος για τον ΙΟΤ ε, που όπως το γνωρίζετε θα αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες για την απορρόφηση των 2 εκατομμυρίων διαρθρωτικών κονδυλίων που θα του δοθούν. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Νταμάτο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Κομισιόν για την παρουσία της, την ε, κυρία Επίτροπο, συγγνώμη. Ε, θα θέσω κάποια ερωτήματα. Η Κομισιόν αποφάσισε να μην προβεί στην διακοπή των προγραμμάτων για την Ισπανία και την Πορτογαλία. Εμεί εκφράζουμε την ικανοποίησή μα, αλλά ταυτόχρονα ε, μα ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι μπορεί να συμβούν κάποια πράγματα στα επόμενα χρόνια για άλλα κράτη-μέλη. Όπω γνωρίζετε, το ΚΟΜ 16 ε, του άρθρου 2003 ε, αναφέρεται ότι θα επαναξεταστεί το εν λόγω άρθρο και η Κομισιόν θα πρέπει να καταρτήσει μια έκθεση που θα υποβάλει το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Σε αυτή την έκθεση ε, μπορεί να συμπεριλαμβάνεται και ένα νομοθετικό, μια νομοθετική πράξη. Ε, για μας ε, θεωρούμε ότι λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της κοινωνικής συγκυρίας που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη θα πρέπει να αντιμετωπιστούν καταλήλως οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι περιφερειακές αρχές. Θα ήθελα να πείσω αν η Κομισιόν έχει παρόμοια πρόθεση. Δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζουμε πως ε, σύμφωνα με τους ε, κανόνες για το πρόγραμμα 2007-2013 και ολοκληρωσίου, οι πληρωμές που έχουν γίνει μέχρι ναι, ναι, το 31 Δεκεμβρίου 2015 μπορούν να μεταφραστούν σε επιστοποιήσεις και αιτήματα μέχρι το 21 Μαρτίου 2017. Σας ρωτώ λοιπόν, δεδομένου ότι έχουμε μελετήσει κάποια στοιχεία πρόχειρα από τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού και αναφέρουν μεγάλη καθυστέρηση στις δαπάνες κάποιων περιφερειών και θα πρέπει να αναφερθώ σε περιφέρειες όπως της Ιταλίας και του Μετζοζόρνου αυτής, εάν σε επαφή με τις κυβερνήσεις ε, ε, είναι σε επαφή με τις κυβερνήσεις Κομισιόν με αυτές τις περιοχές και αν θα πρέπει να ανησυχήσουμε για την απώλεια τυχών κοινοτικών πόρων. Πόροι που ανέκαθεν τονίζαμε ότι σήμερα είναι πολύ πιο απαραίτητοι από το παρελθόν. Σας ερωτώ επίσης, σύμφωνα με την Ιταλική κυβέρνηση, οι αναθέσεις έχουν ήδη γίνει. Και τώρα το μπαλάκι βρίσκεται στο γήπεδο της Κομισιόν οι ε, οποίοι θα πρέπει να προβεί για ορισμού. τους ορισμούς. Μπορεί να δώσει κάποιες πληροφορίες σχετικά, κύριε Επίτροπε. Άκουσα πολλούς συναδέλφους να αναφέρονται στην αλληλεγγύη. Εγώ εκτιμώ ιδιαίτερα αυτές τις δηλώσεις, αλλά να τονίσω όπως χώρες όπως η Ελλάδα και η Ιταλία είναι υποχρεωμένες και μην με παρεξηγήσετε. Το κάνουν για λόγους από ε, τεράστιες ευθύνες να χρησιμοποιούν τους ε, ταμεία, τους ευρωπαϊκούς πόρους που δεν ε, αντιμετωπίζουν τα θέματα τα επίγοντα όπως αυτό της μετανάστευσης. Λοιπόν, κάνω έκκληση προς τους συναδέλφους έτσι ώστε να, ε, να ζητήσουν από τις κυβερνήσεις τους να εφαρμόζουν την αλληλεγγύη σε θέματα μετα, μετανάστευσης και να υλοποιηθούν σε πράξη αυτά τα οποία λένε. Ευχαριστώ. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις από τον πρώτο γύρο από πλευρά συντονιστών. Κυρία Επίτροπε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Εκτιμώ ιδιαίτερα όλες τις παρεμβάσεις και έγιναν κάποιες που επανελήφθησαν και θα ήθελα να απαντήσω σε όλες. Ο κύριος Όλμπριχτ είπε πως ε, αυτή η περιφερειακή πολιτική είχε σχεδιαστεί σύμφωνα με τις συνθήκες για την περιορισμό των ανισοτήτων και πεπισμένη ότι αυτή η πρόκληση υπάρχει ακόμα. Ισχύει. Χρειαζόμαστε αυτή την περιφερειακή πολιτική σήμερα προς ποτέ. Και αυτό με οδηγεί στην δεύτερο ζήτημα περί μη εφαρμογής. Πιστεύω πως αυτά τα οποία πράττουμε σήμερα θα ε, αποτελούν τη βάση για, τις, ε, την επόμενη περιφερειακή πολιτική, την περιφερειακή πολιτική της αύριο. Τώρα, βαζόμενοι στις ε, πληρωμές της Ένωσης, υπάρχει εντύπωση ότι η εφαρμογή αυτών των προγραμμάτων περιφερειακής πολιτικής έχει καθυστερήσει σημαντικά, αλλά η επιλογή προγραμμάτων είναι μια διαδικασία που επιταχύνεται στην Ευρώπη πρέπει να διαφοροποιήσουμε μεταξύ την εφαρμογή προγραμμάτων ε, επιτόπου κάτι το οποίο δαπανούν οι δικαιούχοι και τις πιστοποιημένες δαπάνες που έχουν υποβληθεί ε, στην Κομισιόν μέσω προγραμμάτων. Ε, η επιλογή προγραμμάτων και οι δαπάνες δίνουν μια καλύτερη εικόνα σχετικά με την εφαρμογή της πολιτικής, διότι την εγγύηση για ε, μελλοντικές δαπάνες. Και με ικανοποίηση βλέπω ότι μια αύξηση των επιλεγμένων προγραμμάτων το τέλος του 2015 όπου τα επιλεγμένα προγράμματα ήταν τη τάξη του 250 εκατομμυρίων και τώρα βλέπουμε ότι έχει ανέλθει σημαντικά αυτό το ποσό και η πρωταθλήτρια είναι η Ιρλανδία που έχει ήδη ε, απορροφήσει το 80% των κονδυλίων μόλον ότι οι αρμόδιες αρχές δεν έχουν ακόμα συσταθεί και τη σε λειτουργία. Στο τέλος του 2015 είχαμε ήδη εγκρίνει για στήριξη πάνω από 200.000 επιχειρήσεις και πάνω από 2 εκατομμύρια άτομα εκπαιδεύτηκαν για την, σε, και καταρτίστηκαν για την περαιτέρω αναζήτηση εργασίας. Αυτά είπα και στους υπουργούς την περασμένη εβδομάδα διότι δεν μπορούν να παίζουν παιχνίδια με το μέλλον των πολιτών τους. Έχω και εγώ τις ανησυχίες μου σε τη φορά τις προσωρινές πληρωμές που βάλουν προς την Κομισιόν, διότι υπάρχει αφιβολία σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας, ειδικά στο, ειδικά στο κοινό που δεν γνωρίζει τις ε, ιδιαιτερότητες των πολιτικών μας. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό θα μας πλήξει σημαντικά και πρέπει να το αποφύγουμε. Γνωρίζετε όμως ότι η διαχείριση, η δομή του συστήματος πως είναι, ζητώ από τις αρχές ε, των κρατών μελών, προκειμένου να εργαστούν σκληρά για να επιταχύνουν ε, τις διαδικασίες και οι πληρωμές να καταβληθούν εγκαίρως. Ήμουν σαφής ε, όταν μίλησα στους υπουργούς, στους υπουργούς διότι εμείς είμαστε υπόλογοι και τα κράτη-μέλη εξάλλου είναι υπόλογα. Γι' αυτό θα πρέπει να μας δώσουν κάποιες προβλέψεις. Κάποια κράτη δεν έχουν κατορθώσει να, να απορροφήσουν το 20%. Φυσικά μας ανησυχεί αυτό το γεγονός θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό να ασκήσουμε πίεση προς τα κράτη-μέλη, διότι όταν πρόκειται για εφαρμογή και υλοποίηση, πρόκειται για απόλυτη, απόλυτη ευθύνη των κρατών μελών. Για μας είναι μυστήριο, γιατί αυτός ο ορισμός των ε, θεσμών δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί. Η Κομισιόν τα έχει εγκρίνει και τώρα είναι η ευθύνη των ε, ελεγκτών να ελέγξουν και θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να πετάμε την ευθύνη σαν μπαλάκι από τη μία τον έργο στο άλλο, τον θεσμό στον άλλον. Χαίρομαι που κάποια κράτη έχουν ε, συνάψει αυτές τις συμφωνίες, τις συμβάσεις. Ε, δυστυχώς όμως δεν έχουμε νέα προγράμματα και φυσικά χρειάζεται να εργαστούμε περισσότερο με τα κράτη τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα. Μου είπαν ότι μπορώ να χρησιμοποιήσω και την ε, μητρική μου γλώσσα, αλλά ε, μόνο τα αυτά συνεχίζω στα αγγλικά. Τώρα μιλάτε για τις καθυστερήσεις. Ε, σας πω ότι ο προβλήμα 2017 περιλαμβάνει τις απαραίτητες ε, πληρωμές προκειμένου να τηρήσουμε τις ε, νομικές ε, δεσμεύσεις και δεν θα προβληθούν καθυστερήσεις για το πρόγραμμα 2014-2020 όπως έχει καταδείξει η Κομισιόν υπάρχει μια διάμεση έκθεση αν αυτές οι καθυστερήσεις μόνο ότι είναι χαμηλές θα πρέπει να ε, το ρυθμίσουμε το ζήτημα του προπολισμού Θα πρέπει τα κράτη-μέλη λοιπόν να υποβάλουν προς την Κομισιό προβλέψεις ε, περί των πληρωμών εγκαίρως και ακριβής. Όπως είπα στην ομιλία μου, είμαι έτοιμη να στηρίξω αυτή την πολιτική. Προέρχομαι από μια περιφέρεια όπου η περιφερειακή πολιτική ήταν ένα βασικό στοιχείο των κρατικών επενδύσεων και οι συνάδελφοί μου λένε ότι όλες οι περιφέρειες ε, μπορούν να υποφεληθούν με αυτή την πολιτική και ερώτηση τώρα του κ. Όλμπριχτ δεν είμαι υπέρ της, του διαχωρισμού αυτής της πολιτικής κατά περιφέρεια αλλά νομίζω ότι αυτό θα σήμαινε το τέλος της περιοχής πολιτικής έχω επισκεφτεί 26 κράτη και ε, περιοχές οι οποίες έχουν επωφεληθεί όπως ε, η Βαβαρία ε, θα μεταβώ αύριο στην ε, Λιψία που έχει ανέβει σημαντικά το επίπεδο της λόγω ακριβώς της περιφερειακής πολιτικής. Και κάθε φορά θα πρέπει να τονίζουμε ότι οι περιοχέ του Λουξεμβούργου, το Βέλγιο, την Ολλανδία υποφελούνται από αυτήν την πολιτική. Εντάξει, μιλάμε για διαφορετικό επίπεδο, προκειμένου για θέματα προς την καινοτομία, τις υποδομές, το ε, ε, τομείες στις πλούσιες ε, περιοχές, υποδομές στις φτωχότερες. Έχουμε για την αξιολόγηση εκ των υστέρων 2014-2017. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι για 12 κράτη-μέλη 2007-2013 ήταν ένα πολύ εντατικό πρόγραμμα και είναι φυσιολογικό. θα αφήσουμε στους στους μελετητές, του ιστορικούς να μας πούν κατά πόσον έχουμε χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά αυτό το εργαλείο που είναι διάθεσή μας, αλλά μια που βρισκόμαστε εδώ θα πρέπει να αγωνιστούμε για αυτή την περιφερειακή πολιτική. Και είμαι βεβαία ότι αυτή η πολιτική αφορά όλες τις περιφέρειες, πρέπει να την εξυγχρονίσουμε, να την αναδιαρθώσουμε, να αναδομήσουμε η πολιτική συνοχή θα πρέπει να αφορά τον προγραμματισμό για το μέλλον. Συμμερίζομαι με τις, με τις ανησυχίες σας για τις επιθέσεις που δέχεται αυτή η πολιτική και δεσμεύομαι με τους συναδέλφους μου για την πρόθεση αυτής της πολιτικής διότι θέλουμε να προχωρήσουμε χέρι-χέρι για την ε, ολοκλήρωσή της. Κάθε στιγμή λοιπόν, που έχω την ευκαιρία να μιλήσω με τους συναντέλους μου, τονίζω ότι αυτό είναι πολιτική, δεν είναι ένα οικονομικό εργαλείο μόνο. Είναι η πιο απτή και ορατή πολιτική στην καθημερινή ζωή των πολιτών. Φυσικά η πολιτική συνοχή είναι, ένα θέμα που ενδιαφέρει την, πολιτική Κομισιόν. Ό,τι υπάρχει στο Omnibus σήμερα καθιστά την εφαρμογή της και τη συνεργασία με άλλες πολιτικές πιο αποτελεσματική. Θέλουμε να την ε, διευρύνουμε και με άλλα εργαλεία. Και τελικός στόχος είναι να μην αντικαταστεί η πολιτική στοχή, αλλά να μεγιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις των κοντιλίων μας επιτόπου. Αυτά είναι θέματα που θα πρέπει να τονιστούν. Ε, τώρα για τις καθυστερήσεις μίλησα. Καθυστερήσεις πληρωμές. Όπως είπα, αυτή η πρόταση Omnibus έχει στο στόχο να συνδυάσει τους ε, πόρους από διάφορους οργανισμούς. Έχουμε μια σειρά από εργαλεία και ζητώ από όλα τα κρατη και τα παροτρύνω, ιδιαίτερα της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης που δεν έχουν ε, ε, προγράμματα ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου για θέματα της πολιτικής συνοχής. μπορούμε να λοιπόν, παράσχουμε τεχνική αρρωγή και πιστεύω ότι σημαντικό να συνεργαστούμε και να δούμε στα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ένα σταθερό πλαίσιο για όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων και των πλατφορμών συγχρηματοδότησης. Επόμενο θέμα, αυτό της αλληλεγγύης, που είναι θεμελιώδης σημασία για την Ένωση. δεν είναι μονόδρομος, πρέπει να συνεργαστούμε και κάθε φορά που επισκέφτομαι χώρες οι είναι επιφυλακτικές ε, για, το ζήτημα της μετανάστευσης και της ένταξης των μεταναστών, τους ε, λέω ότι αυτό το θέμα θα επηρεάσει την καθημερινότητα των πολιτών σας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν που στον νέο κανονισμό τώρα υπάρχει, υπάρχει αυτή η προτεραιότητα η οποία παρέχει νομοθετικό πλαίσιο προ όλα τα κρατημέρια να χρησιμοποιήσουν αυτά τα κονδύλια για την ε, ένταξη των ε, μεταναστών. Τώρα λοιπόν καμία χώρα δεν έχει δικαιολογία ότι δεν υπάρχει το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο, αλλά δεν μπορούμε να το επιβάλλουμε να το εφαρμόσουν αυτό το πλαίσιο. Έχω κατά νου αφού εγκρίνεται τον νέο κανονισμό, να σας στείλω με τον συνάδελφο Αβραμόπουλο μια επιστολή προς τα κράτη-μέλη ότι μπορούν να χρησιμοποιούν τώρα τους ευρωπαϊκούς πόρους για τα, τα κέντρα, για τα, ε, ζήτημα υγείας των μεταναστών και να μπορούμε να, να, να ασκήσουμε μια πίεση προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αυτά τα κονδύλια. Όπως είπε η κυρία Νταμάτο, είμαστε αλληλέγγυοι με την Ιταλία και την ε, Ελλάδα και με τη Γερμανία φυσικά που σηκώνουν ένα σημαντικό βάρος. Πρόσφατα ήμουν στην Σουηδία και είδα μερικά πολύ καλά από, παραδείγματα. Δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε σε αυτό το ζήτημα να ε, μας ε, κερδίσει ο λαϊκισμός και τα λαϊκιστικές κορώνες. Είδα να ξεκινάνε, η κατάρτιση για τους δασκάλους από τα σχολεία στην Σουηδία. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τέτοια παραδείγματα και να πολλαπλασιαστούν. Συνάντησα μερικές φορές ε, δημάρχους οι αντιμετωπίζουν διότι μην ξεχνάμε ότι είναι αυτοί οι δήμαρχοι που πρέπει να βρουν άμεσα και κατεπηγόντως λύσεις. Και είχαμε λοιπόν ανταλλαγή απόψεων με αυτούς τους δημάρχους σε αυτή τη συνάντηση και είναι πολύ σημαντικό όπως γνωρίζετε. Διότι κύριε Βεσφάλ ήσασταν εισηγητής ε, για την ε, θεματολόγιο των ε, πόλεων. Είναι λοιπόν σημαντικό να υπάρχουν υψηλής ποιότητας προγράμματα και στο ζήτημα της ένταξης των μεταναστών. Όλα τα κράτη λοιπόν πρέπει να χρησιμοποιούν τουλάχιστον το 5% από το ERDF ε αλλά υπάρχουν κράτη όπως η χώρα από την οποία προέρχομαι που αφιερώνει το 20%. 39 λοιπόν χώρες ε, θα αναλάβουν τη διαχείριση άμεσα. Στην Ισπανία μάλιστα 85 νομίζω. Αλλά αυτό εξαρτάται και από την διοικητική ικανότητα, διότι σε κάποια κράτη η διοίκηση είναι πολύ πιο αδύναμη, δεν έχουν την κατάλληλη εμπειρία για τη χρησιμοποίηση ευρωπαϊκών ενωσιακών πόρων. Αυτή η νέα προτεραιότητα θα πρέπει να την ε, υλοποιήσουν τώρα για το μέλλον της ε, περιφερειακής πολιτικής ε, φυσικά χωρίς να προδιαγράψω μια εξέλιξη για το επόμενο περίοδο θεωρώ ότι θα χρειαστούμε μια πιο ε, ουσιαστική ε, αναθεώρηση. Αυτό είναι ένα, ένα πρόγραμμα το οποίο δεν άλλαξε τα τελευταία 25 χρόνια και δεν μπορούμε να κάνουμε κάποιες ε, κινήσεις σπασμωδικές εδώ και εκεί. Αυτό πιστεύω, αγωνίζομαι γι' αυτό ε, ξεκίνησε μια ζήτηση και στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων από, υπό τη Σλοβακική Προεδρία. Είχαμε μια άτυπη συνεδρία, συζήτηση για το περίοδο μετά το 2020. Κάποια κράτη-μέλη ε, έριξαν την ιδέα για διαφοροποίηση βασιζόμενη στην ιδέα ότι κάποιες ε, δομές διαφέρουν στα κράτη-μέλη και αυτό θα πρέπει να αντανακλάται στο σύστημα λήψη απόφαση. Ε, θα πρέπει να εξετάσουμε λοιπόν αυτή τη διαφοροποίηση και πώς θα προβούμε σε αυτήν. Θεωρώ και εδώ δεσμεύονται και οι συνάδελφοί μου στο απλή της Κομισιόν υπάρχει κάποια, ε, κάποιος δισταγμός ε, αλλά όπου και αν πηγαίνω στις περιφέρειες βλέπω ότι οι δικαιούχοι ζητούν για, ε, κανόνε. για κανόνες ε, Νομίζω πως έχουμε πετύχει κάποια πρόοδο στην εναρμόνιση των κανόνων στο διαφορετικά ταμεία, αλλά σημαντικές ε, διαφορές δημιουργούν ακόμα προβλήματα στους δικαιούχους. Πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια για να περάσουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο, για να έχουμε τους κανόνες για όλα τα ταμεία και την διαχείριση αυτών, αλλά δεν θα είναι εύκολη η συζήτηση. Σκέφτομαι επίσης ε, και τις σημαντικότερες συνέργειες ε, με την χρήση νέων μέσων, όπως είπα, για να ε, μεγιστοποιήσουμε την μόχλευση των κονδύλων του προπολογισμού. Δεν σας κρύβω ότι υπάρχουν προβλήματα. Βλέπω τους εταίρους μου σε αυτόν τον αγώνα, τη μάχη που δίνουμε, ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρξει ένα φόρουμ περί συνοχής και καλύτερα να προχωρήσουμε έγκαιρα κάτι που θα σας επιτρέψει να συζητήσουμε σε βάθος. Τώρα, σε θέμα αφορά την ε, αξιολόγηση ex post, θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τα πρόσφατα ευρήματα τα οποία έχουμε σε αυτό το τομέα και το τι θέλουμε να πετύχουμε. Αυτό είναι πιο σημαντικό με τα χρήματα που έχουμε διάθεσή μας του χρόνου. Λοιπόν, ενδεχομένως να είμαστε σε καλύτερη θέση για την ε, αξιολόγηση των αποτελεσμάτων. Τώρα για την αλλαγή του κλίματος Έχουμε την COP21, θα υπάρξει και COP22. Είναι πολύ σημαντικός πυλώνας για την Ένωση προκειμένου να ε, πετύχει τους στόχους των Παρισίων. Πρόσφατα το Ενεκτικό συνέδριο τόνισε τη συμβολή μας στην προστασία την αλλαγή του κλίματος τώρα, Ισπανία και Πορτογαλία. Ξέρετε πολύ καλά πως δεν ήταν διόλου απλό για μένα να βρεθώ εδώ ενώπιόν σας ε, για να μιλήσω περί θέματος γνωρίζετε πως οι κανονισμοί απαιτούν από την Κομισιόν να υποβάλει αναστολή των διευθυντικών ταμείων εάν το Συμβούλιο αποφασίσει πως το κράτος μέλος δεν έχει αναλάβει δράση για διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος. Αυτή είναι μια νομοθεσία που συμφώνησε και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Και η Κομισιόν φυσικά κατέγραψε τα όσα ελέγχθησαν εδώ, στο Στρασβούργο στην ουσία, ότι ότι υπήρχε μια ομόφωνη θέση με το Ευρωκοινοβούλιο κατά της ε, αναστολής ε, αυτών των προγραμμών προς Ισπανία και Πορτογαλία. Φυσικά λάβουμε υπόψη μας όλα αυτά τα στοιχεία, αλλά γνωρίζετε πως αν τα κρατημέλη δεν ε, λαμβάνουν κάποιες ουσιαστικές δράσεις. Να υπενθυμίσω όμως ότι στο Συμβούλιο κάποια κράτη-μέλη επιχειρηματολόγησαν πως ε, τα αποτελέσματα τα οποία πετύχαμε τώρα προέρχονται από το, το άρθρο 26 γιατί υπήρχε αυτή η απειλή της αναστολής και άσκησε πίεση προ τα κράτη-μέλη για να λάβουν τα μέτρα και να διορθώσουν τον προπολογισμό τους και το έλλειμμα. Το κανονισμό, η Κομισιόν θα πρέπει να προβεί σε μια αξιολόγηση το, μέχρι το 2017 και φυσικά προτιθέμεθα να συντάξουμε μια έκθεση μέχρι τα τέλη του 2017. είναι πολύ νωρίς ε, για να σας πω εάν θα ακολουθήσει και νομοθετική πρόταση Μπορούμε να σκεφτούμε λοιπόν μαζί. Όπως σας είπα, σημασία μεγάλη έχει να είναι όλα έτοιμα. Καταλαβαίνω την κυρία Νταμάτο απόλυτα. Αλλά από την άλλη πλευρά, η άλλη όψη του νομίσματος προέρχεστε από μια περιοχή και γνωρίζετε πολύ καλά ότι έχουμε επενδύσει πολλά χρήματα στο Μετζοζόρνο της Ιταλίας τα τελευταία 40 χρόνια. Και είδαμε ότι δεν έχει αυξηθεί η απασχόληση όσο θα επιθυμούσαμε. Η πολιτική μας δεν μπορεί να λειτουργήσει μεμονωμένα. Έχουμε κάποιες μακροοικονομικές αιρεσιμότητες που θα πρέπει να εφαρμόζονται προκειμένου. Οι επενδύσεις μας θα δημιουργήσουν θέσεις απασχόλησης, ανάπτυξη και βελτίωση του βιωτικού επίπεδου των πληθυσμών. Όταν εγκρίθηκε, εγκρίθηκε ως τελευταία δυνατότητα προσφυγής εάν το κράτος μέλος δεν αναλάμβανε κάποια δράση σχετικά. Το θέμα ε, των εξάντε αιρεσιμότητας είναι ε, πολύ σημαντικό μήμα για να μεγιστοποιήσουμε τις επιπτώσεις ε, των πολιτικών μας επιτόπου. Ξέρετε λοιπόν ότι έχουμε αυτές τις αυτές τις ε, διατάξεις ε, που αφορούν ε, το Μετζοτζόρνο αλλά και το τμήματα της μαλπεριχής της Ισπανίας και το βόρειο τμήμα της Ελλάδος, τη Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει λοιπόν να αποκτηθεί μια στρατηγική για αυτές τις περιοχές. Έχουμε σημαντικά προγράμματα τα οποία εφαρμόζονται τις περιοχές και συμβάλλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών, αλλά θέλουμε να προωθήσουμε ένα νέο πρόγραμμα για να δούμε κατά πόσον όλοι οι παράγοντες που επηρεάζουν την ε, ανάπτυξη των περιοχών μπορούν να συνδυαστούν. Υπάρχουν δύο είδη περιοχών. Όπως το Μετζοζόρνο, όπου επενδύσαμε για πάρα πολλά χρόνια πολλά χρήματα και έχουμε και άλλες περιφέρειες οι οποίες άρχισαν να χρησιμοποιούν ευρωπαϊκούς πόρους εδώ και 10-12 χρόνια και ε, βλέπουμε αποτελέσματα. Βλέπουμε αυτές τις διαφορές ανάμεσα στις δύο περιφέρειες δύο κατηγορίες περιφερειών μάλλον. Ε, η περιφερειακή πολιτική συνοχή ε, καταβάλει κάθε προσπάθεια προς τον... για την ανάπτυξη αυτών των περιοχών, αλλά θα πρέπει όλοι οι εταίροι, περιφερειακοί, τοπικοί, εθνικοί, να συνεργαστούν για την καλύτερη δυνατή χρησιμοποίηση των πόρων ε, συνοχής. Έχω όμως και καλά νέα για το Μέτζο Ζόρνο. Αυτή είναι η πρόγραμμα διοικητικής ενίσχυσης, ενδυνάμωσης έχει αρχίσει να αποφέρει αποτελέσματα και βελτιώνει το θέμα της απλούστευσης των διαδικασιών, ειδικά για τα προγράμματα στο Μετζοτζόρνο. Συνεργαζόμαστε με τις τελικές αρχές για την αύξηση των επενδύσεων στο Μετζοτζόρνο μέσω του Ταμείου και ξέρετε διαξήχθη μια συνάντηση εδώ με όλους τους προέδρους των περιφερειών τον πρόεδρο Κατάινεν και εμού φυσικά και με τα χαράς άκουσα ότι αυτή η συνεδρία αυτή η συνάντηση αυτή τη συνάντηση ακολούθησε μια ιταλική μια τεχνική συνεδρίαση στην Ιταλία και ελπίζω να ε, αποδώσει στις 15 του Δεκεμβρίου θα μεταβώ στην Ιταλία αλλά αυτό το ζήτημα θα αφορά την ελληνική αυτή τη δύσκολη περίοδο πριν από μερικές μέρες λάβαμε έτοιμα για χρησιμοποίηση των, ε, των χρημάτων αλληλεγγύης, χρησιμοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης και να αποσταλούν τα κονδύλια προς την Ιταλία. Ξέρω θα υπάρξει και η ολομέλεια, η οποία θα αφορά τα Ταμείο Αλληλεγγύης. Είναι σημαντικό η περιφερειακή, περιφερειακή αλληλεγγύη να ε, υπάρχει, να ενισχυθεί ιδιαίτερα για τις ε, φτωχότερες περιοχές και τις ε, περιοχές που βρίσκονται, σε μεθοριακές περιοχές. Ήμασταν στην Πορτογαλία, συζητήσαμε γι' αυτό και ο πρόεδρος Γιούνκερ θα καλέσει το Μάρτιο στις Βρυξέλλες εκπροσώπους από τις εξόχως απόκεντρες περιφέρειες για να δείξει την ε, αλληλεγγύη του, την αλληλεγγύη που θα μεταφραστεί και ε, με οικονομικούς όρους. Γνωρίζουμε πολύ καλά ε, τα προβλήματα αυτών των περιφερειών, το δημογραφικό πρόβλημα, τη μεγάλη απόσταση από το κέντρο και όλα αυτά να είστε σίγουροι θα ληφθούν υπόψη στην ανακοίνωσή μας σχετικά με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Μπορείτε λοιπόν να είστε σίγουροι πως θα θέσουμε το θέμα αυτό πολύ ψηλά στον κατάλογο των προτεραιοτήτων. Ο ίδιος ο πρόεδρος Γιούγκερ θα ήθελε να προεδρεύσει σε αυτές τις συναντήσεις. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, όπως συνήθως. Έχω εδώ έναν κατάλογο 7, 8 ε, συναδέλφων που θέλουν να κάνουν ερωτήσεις ή δηλώσεις. Μπορώ να σας δώσω ένα λεπτό στον καθένα, εάν θέλετε να απαντήσει η Επίτροπος. Ε, ναι, κύριε Μόνσκου, ευχαριστώ πολύ, θα προσθέσω και εσάς. Αρχίζουμε με τον κύριο Ντινόλφη. Κυρία Ντινόλφη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Λοιπόν, ε, εγώ είμαι από την περιοχή της Καμπανίας. Ένα από τα μαύρα πρόβατα όταν μιλάμε για κοινοτικούς πόρους. Αυτό που αναρωτιέμαι είναι διότι είναι θετικό το ότι εσείς μας ε, παροτρύνατε να συνεργαστούμε για να βελτιώσουμε την πολιτική συνοχή και την όλη διαδικασία, αλλά έχω ένα ζήτημα πνευματικό θα έλεγα. Γιατί, διότι συνάντησα τον δόκτωρ Μπουτζέλη πριν από ένα μήνα και μετά ε, διάβασα τη δηλώση του που έλεγε ότι η καμπανία είναι ε, το μαύρο πρόβατο όλων των περιφερειών της Ευρώπης και ο δόκτωρ Μπουτζέρη μου είπε ότι όλα πήγαιναν εξαιρετικά, όλα έβαιναν άψογα, ήταν ενθουσιώδης. Όταν του ζήτησα προφορίες σχετικά με τις διοικητικές ικανότητες της περιφέρειας, γιατί και άλλη φορά είχα θέσει αυτό το ερώτημα και γνώριζα ότι οι διοικητικές ικανότητες ήταν ένα από τα βασικά προβλήματα της καμπανίας. Ο, ο Δ. μου είπε ότι δεν έχουν έτσι τα πράγματα και ο δόκτωρ Τόντο, ο οποίος με περιμένει στο γραφείο αυτή τη στιγμή, διαρωτώ με για να βοηθήσουμε την περιοχή και εσείς ως Επίτροπος, ποια, πώς έχει αλήθεια, πώς μπορούμε να επιλύσω ένα πρόβλημα αν έχω δύο ε, αλληλογροθοκοπούμενες πληροφορίες ε, σε ό,τι αφορά την καμπανία. Φαντάζομαι πως ε, ειδικά τα προβλήματα ε, διοικητικής ικανότητας αν έχουν επιληθεί, προβληματα κοινωνικης ικανοτητας αν εχουν επιληθει τοτε η καμπανία δεν θα περιμένει ούτε καν την προθεσμία του 31 Μαρτίου 2017 για να κλείσει τα προγράμματα. Εξάλλου, σε ό,τι αφορά πάντα τη διοικητική ικανότητα της περιφέρειας, είχαμε δήλωση από τον κυβερνήτη της ε, περιφέρειας ότι θα αναλάβει με κοινοτικού πόρους 200.000 άτομα για τη δημόσια ε, διοίκηση. Αυτό το, το συμφώνησε με εσάς τελευταία ερώτηση, ό,τι φορά τη, θέμα, τη μελέτη για τις ε, περιφέρειες της Ρέτζε. εγώ θυμόμουν ότι το Δεκέμβριο θα γίνει αυτή η παρουσίαση. Θα ήθελα να μάθω εάν υπάρχουν και μελέτες ε, ή έγγραφα, κείμενα, εμπιστώσεις που θα παρουσιαστούν ε, για μια διάμεση περίοδο. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν ένα πολύ ιταλικό λεπτό, μακρύ λεπτό. Ε, έχει... Παρακαλώ Ευχαριστώ Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε. Σε σχέση με τα όσα μας είπατε, να περιοριστώ στο να υπενθυμίσω πως ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου εγκρίθηκε, σημαντικό ψήφισμα που αφορά την ιδιαιτερότητα της κατάστασης των νησιωτικών περιοχών. Τα ευρωπαϊκά νησιά μας περίμενα κάτι παραπάνω αυτά τα οποία υπόθηκαν με, και κατά τη διάρκεια τη ε, πρόσφατη συνέντευξή μα. ότι ε, κάποιες μεγαλύτερες ιδιαιτερότητε θα την υπόψη. Υπάρχει ένα μειονέκτημα ε, αυτά τα νησιά και όπω γνωρίζετε, τα νησιά βρίσκονται μονίμως σε μειονεκτική θέση. Ήταν χθε είναι σήμερα και αύριο. Και αυτό τι σημαίνει ότι το, η επιχειρηματικότητα, οι μεταφορές, η ενέργεια, όλα αυτά είναι διαφορετικά, είναι πιο ακριβά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχουν σταθμιμένες πολιτικές για τα νησιωτικές περιφέρειες. Ξεκινώντας και από την ευρωπαϊκή κουλτούρα, τον ε, ορολογία, την πολιτική συνοχή, διότι οι δήμαρχοι μας, σε περιοχές, είναι ε, δήμαρχοι μικρών χωριών. Δεν έχουν καμία δυνατότητα να, να, να δραστηριοποιήσουν κάποιους μηχανισμούς σύνδεσης με την ε, κεντρική κυβέρνηση ή ακόμα και με την Ευρώπη. Είχαμε, είπαμε να οργανωθεί μια υπηρεσία που θα ασχολείται με το ζήτημα αυτό και εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι κατεπήγον. Φυσικά θα ζητήσουμε για τα ταμεία και για το ψήφισμα που εμείς έχουμε παρουσιάσει σχετικά με τον σεισμό. Χαίρομαι που στις 15 Δεκέμβρη θα μεταβείτε στην Ιταλία και να μην ξεχνάμε ε, να ε, μην ξεχάσουμε ε, τα θύματα αυτών των καταστροφικών σεισμών. Κυρία Μπρέσο, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σε αυτή την Επιτροπή γίνομαι εμπειρογνώμων σιγά-σιγά. Και σας ερωτώ, επειδή είναι προφανώς, προφανές ότι το όργανο δεύσει γίνεται ο ανταγωνιστής για πώς ε, μπορούμε εμείς να υποφελθούμε από την ικανότητα συνεργασίας ε, των δύο ταμείων. Δηλαδή, δεν ε, θεωρείται ότι θα μπορούσε να γίνει ένα συμβουλευτικό όργανο σε εθνικό επίπεδο που θα βοηθάει τις περιφέρειες στο να χρησιμοποιούν από κοινού τα δύο αυτά μέσα, δηλαδή το Ευρωπαϊκό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Ταμείο να γίνει ε, αρρωγός του πολιτικής συνοχής και όχι αντίπαλος. Τώρα ένα από τα προβλήματα για την καθυστέρηση της ανάθεσης των πόρων στην περιφέρεια είναι ότι όταν τα προγράμματα ε, υποβάλλονται, τότε αρχίζουν οι καταβολές. Θα πρέπει να γίνει μια καλύτερη κλιμάκωση αυτής της διαδικασίας ε, ήδη με την υποβολή να υπάρχει προχρηματοδότηση για την μελλοντική το μελλοντικό πρόγραμμα, μελλοντική υποβολή από τη στιγμή φυσικά όπου οι, οι γραμμές της μελλοντικού προγραμματισμού θα έχουν ξεκινήσει ένα χρόνο πριν, παραδείγματο χάρη. Γιατί να μην έχουμε κάποια κονδύλια αυτή εξ αρχή, τα οποία θα ε, χορηγούνται για την επόμενη υποβολή του προγράμματο. Το γεγονός είναι ότι αρχίζουμε να προγραμματίζουμε όταν φτάσουν τα χρήματα, ενώ θα πρέπει τα προγράμματα να είναι έτοιμα. Ευχαριστώ την Τζουφρή το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστούμε την κυρία Επίτροπο την οποία και ε, όλοι τις αναγνωρίζουμε ότι συνεχίζεται αυτός ο διάλογος μεταξύ ημών και της ε, Επιτρόπου. Ακούσαμε νέες ειδήσει, ευχάριστες για τις εξελίξεις στο Μιτζοζόρνο, και σε σχέση με αυτή τη δημοσίευση. Βλέπουμε ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια του ότι ένα ευρώ που επενδύεται στην πολιτική συνοχή γίνονται μετά από μερικά χρόνια 2,74 και η αντίληψη όμως στην Ιταλία δεν είναι αυτή, ειδικά στις περιοχές του Μέτζο Τζόρνου, όπου ζουν σε, ένα φοβερό χάσμα μεταξύ της υπόλοιπης Ιταλίας. Θα ήθελα να μιλήσω για την τήρηση των κανόνων, κάτι το οποίο συζητήθηκε πολύ τα τελευταίες εβδομάδες, ειδικά στο πλαίσιο των συζητήσεων που έγινε για την Πορτογαλία. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν στα προγράμματα της Κομισιόν να συνδυάσουν τη χρήση των ε, διαφορετικών ταμείων στην, ε, και στην τήρηση του κράτους δικαίου αλλά και της αλληλεγγύης. Βλέπουμε ότι η αλληλεγγύη ακούγεται συνεχώς σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μιλάμε ιδιαίτερα στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής που θα πρέπει να είναι το ε, κατεξοχήν όργανο. Η Ιταλία είναι κάποια χώρα η οποία ευνοείται τα μάλα από την πολιτική αυτή. Τώρα, η ερώτηση έχει εξή, γιατί τα διευθυντικά ταμεία δεν διακόπτονται στα κράτη όπου η αλληλεγγύη δεν εκδηλώνεται, ενώ διακόπτονται ή αναστέλλονται ή απειλούν να ανασταλούν σε χωρε οι οποίες αντιμετωπίζουν τεράστια οικονομικά προβλήματα. Όλα αυτά προκαλούν μια αμφιβολία και μια επιφύλαξη από πλευρά ε, των πολιτών. Λοιπόν, το ερώτημα είναι να δουλέψουμε περισσότερο σχετικά με την σύλληψη των προγραμμάτων. Η Κομισιόν καταβάλει προσπάθειες, αλλά η πολιτική συνοχή όταν επιτυχάνεται δυστυχώς δεν γίνεται γνωστή, δεν γνωστοποιείται. Και αυτή η τεράστια διαφορά που υπάρχει για μια χώρα όπως την Ιταλία που είναι πραγματικά ανυπόφορη. Κυρία Ροντρίγκης, προσπάθησα να τηρήσω το λεπτό μου. Ήθελα να μιλήσω πορτογαλικά, αλλά βλέπω πως σήμερα δεν έχω αυτή τη δυνατότητα, οπότε θα τα πω αγγλικά. Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους, την Επιτροπή μας εδώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που προσπαθεί να μην επιβληθούν οι κυρώσεις ε, στη χώρα μου και στην Ισπανία. Χρειάζεται να επανεξετάσουμε το άρθρο 23. Ε, εσείς ε, τι σκοπεύετε να κάνετε για το θέμα αυτό. Έχω και δύο ερωτήσεις, αλλά δεν μου φτάνει χρόνος, οπότε θα κάνω μόνο τη μία. Έχετε κάποια πρόταση για συγκεκριμένα μέτρα ε, αντιμετώπισης του προβλήματος ε, της ανταγωνιστικότητας σε αυτές τις εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ο κύριος Γιούνκερ έχει τοποθετηθεί για την ε, πολιτική συνοχή. Εσείς έχετε κάποια ε, πρόταση για το πώς μπορούν να λυθούν αυτά τα προβλήματα στις ε, εξόχως απόκεντρες περιοχές. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ρούις έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω τη γλώσσα μου. Όχι, συγγνώμη, δεν υπάρχει διερμηνία στα πορτογαλικά, δεν μπορείτε. do meu vizinho espanhol. É também uma assimetria, Sra. Presidente. Συγγνώμη κύριε Ρουίς, δυστυχώς δεν υπάρχει διερμηνία από τα πορτογαλικά. Προσπαθήστε στα γαλλικά, στα αγγλικά, σε κάποια άλλη γλώσσα. Όχι, δεν, δεν επιθυμώ να μιλήσω γαλλικά. Θα ήθελα να μιλήσω πορτογαλικά, αλλά γι' αυτό... Δεν θέλω να μιλήσω γαλλικά, θα ήθελα να μιλήσω πορτογαλικά, γι' αυτό λοιπόν θα αφήσω την ερώτησή μου για κάποια άλλη στιγμή. Στην Πορτογαλία επιθυμούμε, ξέρετε, να μιλάμε τη μητρική μας γλώσσα και αυτό θα πράξω κιόλα και θα το κάνω στο μέλλον. Yes, I'm... Μάλιστα, συμφωνώ απόλυτα με αυτό. Έχετε κάθε δικαίωμα να μιλήσετε τη γλώσσα σας. Δυστυχώς όμως σήμερα δεν υπάρχει ε, διερμηνία σε όλες τις γλώσσες. Δεν είναι μόνο η δική σας, υπάρχει, ε, υπάρχουν και άλλες γλώσσες που δεν έχουν διερμηνία, ούτε τα ρουμάνικα έχουν διερμηνία. Αυτό είναι το πρόβλημα, ξέρετε, που έχουμε καμιά φορά στο Κοινοβούλιο. Ε, κύριε Χέντμαν, έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επίτροπο που ήρθε στην Επιτροπή μας. Δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαν οι άλλοι συνάδελφοι. Συμφωνώ απόλυτα με την ε, κυρία Επίτροπο. Θα ήθελα να πω μόνο. Υπάρχουν καθυστερήσεις στην πολιτική συνοχής. Ταυτόχρονα όμως υπάρχουν και διαφορές ως προς τον αριθμό των ε, συμβάσεων που υπογράφονται, των πιστοποιήσεων ε, για ορισμένες περιφέρειες. Σε ορισμένες περιφέρειες είναι ταχύτατη η ρυθμή ε, των υπογραφών αυτών των συμβάσεων και μάλιστα υπήρχε συσσόρευση σε κάποιες από αυτές τις περιφέρειες πληρωμών. Πώς θα μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση και γιατί υπάρχουν τέτοιες καθυστερήσεις. Είναι μια πολύ απλή ερώτηση, αλλά μου φαίνεται πως δεν θέλει ή δεν μπορεί κανείς να δώσει τα τελευταία δύο χρόνια μια απάντηση. Τώρα, σε ό,τι αφορά την ε, υλοποίηση έργων, προγραμμάτων, πιστοποιήσεων, υπογραφή συμβάσεων, υπάρχει τεράστια γραφειοκρατία κατά την αξιολόγηση έργων, κατά την ε, υλοποίησή τους, κατά την διευθέτηση λογαριασμών, την παρακολούθηση των έργων αυτών. Αυτό απαιτεί χρόνο. Χρόνος ε, ο οποίος αφαιρείται από εμάς, χρόνο τον οποίο θα έπρεπε να αφιερώνουμε στην συνέχιση της πολιτικής, στην επιτάχυνση των προσπαθειών μας. Ε, κυρία Επίτροπε, έχετε την ευκαιρία να γραφτείτε στις χρυσές σελίδες αυτής της ε, Ένωσης, εάν επιβάλλετε ελέγχους ελέγχου σε περιφέρειες όπου παρατηρείται πάρα πολύ μεγάλη γραφειοκρατία. Εάν εσείς ε, βάζατε την ε, αρχή για να γίνουν αυτοί οι έλεγχοι, τότε θα μπορούσαμε να δούμε τι γίνεται σε κάθε κράτος μέλος, ποια πράγματα πρέπει να αλλάξουν, πρέπει να καταργηθούν, ποιες απαιτήσει πρέπει να ε, χαλαρώσουν. Αυτό πιστεύω θα έδινε το πράσινο φως ε, σε όλους τους υπόλοιπους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θα έδινε το πράσινο φως για να είμαστε περισσότερο ευέλικτοι, για να εφαρμόσουμε την πολιτική και αυτή η πολιτική να αποδώσει καρπούς. Τέλος, έχουμε προσπαθήσει πολλές φορές να πείσουμε τους αυτούς μας ότι η πολιτική συνοχή είναι αν όχι η πιο σημαντική η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τις σημαντικότερες έστω. Και προσπαθούμε να πείσουμε τους αυτούς μας πάλι ότι αυτό αφορά όλους τους πολίτες της Ένωσης. Και το επαναλαμβάνουμε. Επαναλαμβάνουμε επίσης ε, συχνά ότι η πολιτική συνοχή είναι ο τράγος, ότι ε, προσπαθούμε μέσω αυτής να λύσουμε όλα μας τα υπόλοιπα προβλήματα. Όμως, όταν υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα, δεν θα έπρεπε να αναλογιστούμε γιατί υπάρχουν αυτές οι καθυστερήσεις. Γιατί μήπως επειδή δεν προωθούμε τα ε, ταμεία συνοχής, μήπως επειδή δεν κάνουμε καλά τη δουλειά μας. Και εδώ έχετε κι άλλη μια ευκαιρία να γραφτείτε στις ε, χρυσές σελίδες της ιστορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν κατευθυντήριες γραμμές για τα πάντα. Και όλα περνάνε μέσα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, αφορούν την προώθηση αυτών των ε, ταμείων. Ίσως αν τις ακολουθούσαμε να ήταν καλύτερα τα πράγματα, αλλά να σας πω εγώ ότι ο ε, απλός πολίτης δεν τα βλέπει αυτά τα αποτελέσματα της πολιτικής συνοχής. Όμως είναι ορατά αρκεί να ξέρει κανείς που να κοιτάξει. Πρέπει λοιπόν να ε, ορίσουμε εκ νέου την ε, συνοχή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα είχα πολλά να σας πω, αλλά δυστυχώς δεν έχω πολύ χρόνο στη διάθεσή μου. Ευχαριστούμε που αφιερώνετε λίγο χρόνο για να συζητήσουμε μαζί ε, το θέμα της ε, περιφερειακής πολιτικής και κυρίως ε, για το ότι επιβεβαιώσατε την αποφασιστικότητά σας και την αφοσίωσή σας ώστε αυτή η πολιτική της κοινωνικής συνοχής να εφαρμόζεται στο δυνατό καλύτερα σε ενωσιακό επίπεδο. Είτε το θέλουμε είτε όχι ο στόχος ήταν η μείωση των ανισοτήτων μεταξύ των ε, ε, πολιτών. Ε, τα αποτελέσματα είναι απτά σήμερα. Έχουμε επιτύχει. Να σας πω ένα παράδειγμα θετικό των διαμερισμάτων της, των υπερποντίων της Γαλλίας, των άκρος περιφερειακών περιοχών. Μπορούμε να δούμε πλέον τι έχει γίνει. Είχα πάει και στη Μαδέρα προς ε, προσφάτως και είδαμε τι ακριβώς έγινε. Ε, νομίζω ότι πραγματικά ενισχύσαμε τους πολίτες μας ώστε να μπορέσουν ε, να ζήσουν καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω να συνεχίσετε με την ίδια θέληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να σας ζητήσω, κυρία Επίτροπε, να απαντήσετε όσο το δυνατόν συντομότερα, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πρέπει να μιλήσω Ιταλικά με όλους τους ε, συναδέλφους που πήραν το λόγο στα Ιταλικά, αλλά θα τα πω στα Αγγλικά. Δεν είναι αλήθεια αυτό που είπατε. Εμείς ε, δεν καταλογίζουμε τίποτε σε κανέναν ε, δάκτυλο δεικνύοντάς τον, αλλά ε, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβαίνει. Μας είπαν από τη Γενική Διεύθυνση ότι η Καλαβρία, η Καμπανία και η Σικελία δεν θα ολοκληρώσουν τα επιχειρησιακά προγράμματα μέχρι την προθεσμία. Εγώ είχα πάει στην καμπανία ε, της Ιταλίας, ε, γνώρισα όλους τους ε, αρμοδίους φορείς, η καμπανία ήταν η τελευταία, αλλά ήταν και η δυσκολότερη ως προς την προθεσμία. Είναι γεγονός ότι η διοικητική ικανότητα είναι προβληματική εκεί, αλλά έχουμε αυτό το πλαίσιο καλύτερης εφαρμογής που έχει κάποια αποτελέσματα στην Ιταλία και όπως είπα υπάρχει αυτό το πρόβλημα της διοικητικής ικανότητας γενικότερα για την Ιταλία. Ε, ε, θα γνωρίσω μάλιστα ε, τον αναπληρωτή πρωθυπουργό στη Ρώμη και θα μιλήσουμε μακροσκελώς για αυτό το θέμα κατά την επίσκεψή μου στην Ιταλία σε δύο εβδομάδες από τώρα. Οπότε σε κάθε περίπτωση σας ενθαρρύνω να μεταφέρετε το μήνυμά μας ότι μαζί σας είμαστε και είμαστε έτοιμοι να ε, κάνουμε όλες τις προσπάθειες και σε τεχνική αρρωγή και σε εμπειρογνωμοσύνη για να καλύψουμε το χάσμα. Ε, χάρηκα πάρα πολύ που εγγενιάσαμε το σιδηρόδρομο μεταξύ Μπάρι και Νάπολης. Ε, είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και η Ιταλία νομίζω ότι είναι το σημαντικότερο παράδειγμα ε, ότι δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη, αλλά και εντός των κρατών μελών υπάρχουν τεράστιες ανισότητες και αυτός είναι ένας ακόμη λόγος για τον οποίο πρέπει να ε, αγωνιστούμε για αυτήν την περιφερειακή πολιτική. Υπάρχουν πολλά επιτεύγματα, αλλά υπάρχουν και κάποιες περιφέρειες οι οποίες δεν τα πηγαίνουν καλά. Ε, πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και αν υπάρχει αυτή η ισορροπία, ε, αν δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία σημαίνει ότι δεν έχουμε κάνει αρκετά ε, σε επίπεδο εθνικών αρχών. Έχετε ένα πάρα πολύ Ιρλανδικό όνομα, ένα πολύ Ρουμανικό όνομα, κύριε ε, Τσίκου. Είχαμε αυτή τη συζήτηση, είχαμε συζητήσει όπως είπαμε ε, και μαζί, να αντιμετωπίσουμε τις ιδιαιτερότητες των νησιών ε, των νησιωτικών περιοχών και κάνουμε κάποιες αλλαγές τώρα στο πλαίσιο της Γενικής Διεύθυνσης ε, Περιφερειακής ε, Ανάπτυξης και προσπαθούμε να υπάρξει ένα πλαίσιο στενή συνεργασίας για να αντιμετωπίσουμε το θέμα των νησιωτικών περιοχών με τη χρήση των καλύτερων πρακτικών, την αντιμετώπιση των προβλημάτων, τις καλύτερες λύσεις κλπ. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι κατόπιν αιτήματος των κρατών μελών ε, ε, δημιουργήσαμε αυτό το... Ε, ούτε αυτό το, αυτό το, αυτήν την προσπάθεια είναι στο, στη ε, συνθήκη της χώρας σας με την Ευρωπαϊκή ε, Ένωση. Ούτε η Ελλάδα, ε, ούτε η Ιταλία θέλησαν να είναι τμήμα του ιδίου προγράμματος, παρά το γεγονός ότι έχουν νησιά. Καταλαβαίνω όμως πάρα πολύ καλά τι είπατε. Τα νησιά πρέπει να την χάνουν διαφορετικής μεταχείρισης και όπως είπα σε κάθε ε, συζήτηση υπάρχει κάποιος ο οποίος ασχολείται με τα ε, νησιά, όπου υπάρχουν νησιά ε, στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οπότε βεβαίως θα λάβουμε υπόψη αυτήν την ιδέα για την ενιαία θηρίδα. αλλά θα πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα. Κυρία ε, Ροντρίγκε, νομίζω ότι αυτός ο πυλώνας ε, είναι ένας από του πιο σημαντικού ε, η προσβασιμότητα στον τομέα των μεταφορών, όπως επίσης και η αύξηση της απασχόλησης είναι πολύ σημαντική. Όσον αφορά το Ταμείο Αλληλεγγύης, όπως είπα, αύριο στην Ολομέλεια θα το συζητήσουμε όμως αυτό που θα ήθελα να σας πω εδώ επειδή είναι τόσο πολύ ε, οι Ιταλοί, ε, είμαστε σε πλήρη αλληλεγγύη μαζί τους ε, και με τις ε, ε, αρμόδιες αρχές μετά από τον σεισμό το Ταμείο Αλληλεγγύης είναι ένα από τα ισχυρότερα συμβολά μας ως προς την αλληλεγγύη που επιδεικνύουμε όταν υπάρχει ανάγκη. Η Ιταλία ήταν ο μεγαλύτερος ε, δικαιούχος αυτού του Ταμείου από την ε, ε, ίδρυσή του με 1,3 δισεκατομμύρια που κινητοποιήθηκαν υπέρ της μέχρι τώρα. Ναι, αυτό φυσικά δεν είναι ευχάριστο αλλά σε σχέση με, την, τον τελευταίο σεισμό ε, έκανε αίτηση η Ιταλία για την αρρωγή από το Ταμείο Αλληλεγγύη. Λάβαμε τον Οκτώβριο την αίτηση Τώρα ε, προσπαθούμε να ε, το επεξεργαστούμε για να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τις εργασίες οικοδόμησης στη χώρα. Επίσης, ε, είμαστε σε έντονο διάλογο και εξετάζουμε από κοινού με τις Ιταλικές Αρχές την δυνατότητα χρησιμοποίησης ε, του μαθηματικού στόχου 416 ε, για την ε, κοινωνική ενσωμάτωση όπως επίσης και την αντιμετώπιση των προβλημάτων των σεισμών στο περιβάλλον. Μου λένε επίσης ότι υπάρχει ένα πρόβλημα με το χρόνο και ότι πρέπει να ολοκληρώσω, αλλά να ξέρετε ε, ότι είμαστε μαζί με τον Ιταλικό λαό σε, αυτό το δύσκολο, σε αυτή τη δύσκολη ε, συγκυρία. Ε, όπως είπα, πρέπει κύριε Πρέστο να είμαστε να συνεργαστούμε δεν είναι θέμα ανταγωνισμού το οικονομικό μέσο ε, δεν ε, μπορώ να σας πω τίποτε άλλο εκτός από το ότι υπάρχει ένας νέος κανονισμός, το Omnibus που εγκρίθηκε ε, για... υπάρχει και ένας ε, ειδικό απεσταλμένος που προβλέπεται στο πλαίσιο του κανονισμού αυτού για να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει συνεργασία ε, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει ένα δίκτυο σε πολλά κράτη-μέλη δεν γνωρίζουμε πού να στραφούμε στο Υπουργείο ε, Οικονομικών ή σε κάποιο άλλο Υπουργείο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να έχουμε με κάποιον ο οποίος ασχολείται ε, με ε, τα θέματα αυτά, τα περιφερειακά και νομίζω ειδικότερα στην περίπτωση αυτού του οικονομικού μέσου είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Έχετε δίκιο πάντως ε, ότι ένα από τα ζητήματα για τα οποία πρέπει να συνεργαστούμε είναι ο καλύτερος τρόπος ε, να υπάρξει μια ομαλή μετάβαση από τη μία περίοδο στην άλλη και πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι εν Αυτές Αυτή είναι μία από τις ιδέες μας, να υπάρχει ένα δίκτυο μεταξύ κρατών μελών και Ευρωπαϊκής Επιτροπής εντός ε, της αντιπροσωπείας για να υπάρχει μία σαφής εικόνα επιτόπου για το τι πρέπει να γίνει και τι μπορεί να γίνει. Και Όσον αφορά ε, στο τελευταίο ερώτημα, για την εφαρμογή. Κύριε Χένμαν, αυτή η εντύπωση που έχετε ότι η εφαρμογή είναι πολύ βραδία, 120 δισεκατομμύρια είχαμε γκρίνει για την προγραμματική περίοδο. Είναι πολλά χρήματα από τα 400 δις. Πάντως αυτό δεν αντανακλάται γιατί τα κράτη-μέλη δεν υπέβαλαν ε, τις ε, πιστοποιημένες ενδιάμεσες πληρωμές ε, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με ρωτήσατε γιατί. Κοιτάξτε, εγώ δεν έχω σαφή απάντηση να σας δώσω και για μένα αποτελεί μυστήριο για ποιο λόγο δεν πιστοποιούν συντομότερα από τη στιγμή που δεν έχουν ε, αυτές τις πιστοποιήσεις, δεν ε, έχουν τα τιμολόγια και δεν μπορούν να πληρώσουν. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχουν αυτά ε, τα όργανα ώστε να αρχίσει η πραγματική εφαρμογή. Νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και θέσατε επίσης ένα ακόμη σημαντικό ζήτημα της γραφειοκρατίας γιατί εδώ ε, δουλεύουμε για την απλοποίηση του κανονισμού, ε, γιατί πολλά κράτη-μέλη όλο και προσθέτουν κάτι Ε, κάποιοι δήμαρχοι από τη δική μου τη χώρα μου είπαν ότι δεν μπορούν ε, για αυτό το πρόγραμμα ενεργειακής αποδοτικότητας, δεν, μπορούν να κάνουν αίτηση. Είναι ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα γιατί πρέπει να δείξουν ε, ότι μεταξύ της δεκαετίας του 70 και του 90 οικοδομήθηκαν αυτά τα κτίρια. Οπότε αντί να ε, συγκεντρωθούν στη δουλειά, πρέπει να βρουν ε, χαρτούρα για να δικαιολογήσουν το αίτημά τους. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ε, τι να σας πω, ε, δηλαδή αν κάποιο οικοδόμημα χρονολογείται από το 1920 δεν μπορεί να είναι επιλέξιμο ή αν είναι του 91, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Ε, είναι πάρα πολύ περίεργο και σε μερικά κράτη-μέλη βρίσκω πολλούς τέτοιους περιορισμούς που δεν είναι απαιτήσει Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί μόνο στον κανονισμό για τι κοινέ διατάξει υπάρχει 600 600 σελίδες. Γιατί χρειάζονται τόσες πολλές ε, σελίδες και τόσες πολλές απαιτήσει. Νομίζω ότι είναι ήδη αρκετά περίπλοκη η κατάσταση. Ε, όχι επειδή θέλουμε να είμαστε περίπλοκοι, αλλά γιατί πρέπει να βρούμε την ισορροπία μεταξύ της απλοποίησης, που είναι το βασικό ζήτημα εδώ πέρα ε, στην Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης, και την επόμενη εβδομάδα θα μιλήσουμε για τη λογοδοσία, για το πώς ε, δαπανώνται τα κονδύλια και θα πρέπει να βρεθεί βεβαίω ένας, ε, ε, μια ισορροπία και τα κράτη-μέλη πρέπει να καθυσυχαστούν ότι τα χρήματα δαπανώνται με κάποια διαφάνεια. Από την άλλη, πολλές φορές δεν μπορούμε να συσβιβαστούμε γιατί οι πολιτικές μας στοχεύουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και μερικές φορές γίνονται γραφειοκρατικοί. Παρ' όλα αυτά δεν φταίμε πάντοτε εμείς. Ε, είναι και τα κράτη-μέλη μερικές φορές που δεν κάνουν τη δουλειά τους στο πλαίσιο της απλοποίησης. Τώρα έχουμε ας πούμε τη e-cohesion, ε, ένα σύστημα ε, ηλεκτρονικής απλοποίησης. Αυτή τη στιγμή θα έχει εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτή, αυτό το Omnibus θα ε, γυρίσει πάλι σε εσά ε, για να, γνωρίσει, να το γνωρίσουν τα κράτη-μέλη και να δείτε τις νέες ε, δυνατότητες απλοποίησης των διαδικασιών. Ευχαριστώ λοιπόν πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήμουν εδώ. Πάντοτε θέλω να ανταλλάσσω απόψεις μαζί σας για τέτοιου είδους θέματα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο για μένα και με βοηθά πάρα πολύ να συνεχίσω και να αγωνίζομαι για την πολιτική αυτή. Αυτός θα είναι ο στόχος μας ε, για την επόμενη χρονιά, γιατί θα είναι μια κρίσιμη χρονιά και αν δεν σας δω μέχρι το τέλος της χρονιάς, ε, θα ήθελα να σας ευχηθώ ε, ό,τι καλύτερο. Ελπίζω να ξαναβρεθούμε στις αρχές της χρονιάς με πολλά καλύτερα νέα, γιατί ελπίζουμε ότι μέχρι το τέλος του Δεκεμβρίου του τρέχοντος ε, πολλές από αυτές τις εκ των προτέρων ερεσιμότητες θα έχουν εκπληρωθεί και επίσης μπορούμε να ε, λάβουμε και ε, όλα αυτά τα δικαιολογητικά για τις πληρωμές για να μπορούμε να έχουμε και από εσά πάρα πολύ καλά νέα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κυρία Επίτροπε. Εκ μέρους όλων των μέλων της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης είστε ευπρόσδεκτοι όποτε θέλετε να έρθετε σε εμά. Και θα ήθελα εδώ να ευχαριστήσω τους διερμηνείς για την κατανόηση που έδειξαν. Διακόπτουμε λοιπόν τη συνεδρίαση μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Ευχαριστώ.